Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το απογευματινό τμήμα της συνεδρίασης. Θα συζητήσουμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα στην Ιρλανδία και πιο συγκεκριμένα ένα πρόγραμμα που συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με το Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία. Έχουμε εδώ διάφορους ομιλητές αυτούς που ασχολούνται με την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. Θα ακούσουμε τον Πατ Κόργαν, που είναι επικεφαλής των ειδικών, του ειδικού φορέα για τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που ασχολείται με τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Περιφερικής Πολιτικής και ο Ρούνι είναι πρόεδρος του Διεθνούς Ταμείου για την Ιρλανδία και παρευθύνσεις θα σας ακούσουμε. Πατ, ξεκίνα. Είναι εκτός μικροφώνου, δυστυχώς δεν ακούμε τον ομιλητή. Δεν ακούνε οι διερμηνείς τον ομιλητή. Okay. Thank you very much, Chair. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα, θα γνωρίζετε το ειρηνιστικό πρόγραμμα της, και την ειρηνιστική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία διότι ήσασταν επίτροπος πλήν και έχετε επισκεφθεί επανειλημμένα την Ιρλανδία. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε για να μιλήσουμε στην Επιτροπή σας για να αναφερθούμε στο έργο μας. Εν συντομία, είμαι επικεφαλής μιας οργάνωσης Special EU Programs Body αποκαλείται, ειδικό φορέ του προγράμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωσης βασίζεται στη Συμφωνία του Μπέλφαστ της Μεγάλης Παρασκευής ε, του 1998, συνήφθη μετά την κατάπαυση του πυρός, δημιουργήθηκε από τη Βρετανική και την Ελληνική Κυβέρνηση και είναι ένας από τους έξι εφαρμοστικούς φορείς που εμπλέκονται σε ένα φάσμα δραστηριοτήτων συνεργασίας σε διασυνοριακό επίπεδο μεταξύ Δημοκρατής Ιρλανδίας και Βορείου Ιρλανδίας. Είμαστε υπεύθυνοι για τη χρηματοδότηση για τον χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσης, το Interreg και για, την, και για το PIS, για την ειρήνη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ερχόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι είναι το σπίτι των ενευτικών προγραμμάτων Κοινοβούλιο του 1995 με πρωτοβουλία τριών ευρωβουλευτών τότε της Βορειοελλανδίας που μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβαν την πρωτοβουλία, δημιούργησαν την πρώτη πρωτοβουλία για το ειρηνευτικό πρόγραμμα και νομίζω ότι είναι σωστό και δίκαιο που είμαστε εδώ για να αποτίσουμε φόρο τιμή στο ρόλο που το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε ε, με τη σειρά με την πάω των ετών για την ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία. Και εντωμεταξύ είχαμε πρωτοβουλίε από την Μπάρμπαλα Ντεμπρούν που ανήκε στην επιτροπή αυτή που έκανε παρέμβαση και συνέταξε έκθεση που συμπλήρωσε και την έκθεση και το έργο που ε, έγινε από την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το Ειρηνευτικό Πρόγραμμα και ε, εξετίμησαν τα μάλα τα επιτευθέντα του ειρηνευτικού προγράμματος οι δύο εκθέσεις. Ε, θα ήθελα ακροθυγώς να αναφερθώ στις αρχικές φάσεις, τις πρώτες μέρες. Όπως είπα, ανταπόκριση σε πρωτοβουλή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1995 εφαρμόστηκε το πρώτο σημαντικό ειρηνευτικό πρόγραμμα. Τότε το καθήκον ήταν να αντιμετωπιστεί η κληρονομιά της σύγκρουσης στην περιοχή, στην Βόρεια Ιρλανδία και στις διάφορες κομιτείες των, της παραμεθόριας. Υπήρχαν διάφορα προβλήματα να αντιμετωπιστούν τότε. Είχαμε πολύ σημαντική ειρηνευτική διαδικασία που ε, λάμβανε χώρα, εκφραζόταν από τις δύο κυβερνήσεις και τους βασικούς εμπλεκομένους φορείς στη Βόρεια Ιρλανδία και στην Ιρλανδία, αλλά τα ειρηνευτικά προγράμματα όταν εφαρμόστηκαν έγιναν ειρηνευτική διαδικασία του λαού έγινε η ρευτική διαδικασία, η επιτόπια, η ρευτική διαδικασία στους δρόμους. Συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου σε διάφορες ειρηνευτικές διαδικασίες. Το δεύτερο πρόγραμμα ξεκίνησε το 2000 και βασίστηκε στην επιτεφίσα μέχρι τότε πρόοδο. Και τώρα είμαστε στο τρίτο πρόγραμμα, το οποίο προσπαθεί να βασιστεί στην επιτεφίσα πρόοδο, αλλά να αντιμετωπίσει τα προβλήματα εμπιστοσύνης που υπάρχουν ακόμα ε, όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των κοινοτήτων στη Βόρεια Ιρλανδία. Όσον αφορά το μέλλον, προσβλέπουμε στην ε, συνέχεια των εργασιών και είναι σωστό να πούμε ότι φύγαμε από τη δυσκολότατη αρχική περίοδο και φτάσαμε στα, στις διαδικασίες που εξακολουθούν να είναι πολύ δύσκολα όσον αφορά την εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινοτήτων και παρόλο που πετέχσαν πολλά, πολλά απομένουν να γίνουν, πάρα πολλά. Αν δείτε το χάρτη, θα δείτε την περιοχή που καλύπτουμε. Έχουμε γαλάζια όλη τη Βόρεια Ιρλανδία και στα κόκκινα έχουμε τις έξι παραμεθόριες κομιτείες της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Συνολικός πληθυσμός σε αυτή την περιοχή 1,6 εκατομμύρια στην Βόρεια Ιρλανδία, περίπου 500.000 ε, στις παραμεθόριες κομιτείες της Ιρλανδίας και όπως σας είπα ε, τα προγράμματα PIS επί σειρά ετών ε, ήταν σημαντικό κομμάτι της ειρηνευτικής διαδικασίας και εγώ θα έλεγα ότι είναι η ειρηνευτική διαδικασία του λαού. Πάρα πολλά προγράμματα, πάνω από 15.000 το πρώτο πρόγραμμα και πάνω από 7.000 προγράμματα μέσω του PIS 2 με πάνω από 995 εκατομμύρια ευρώ και με το παρόν πρόγραμμα που είναι πιο μικρό στρατηγικό εστιασμένο πρόγραμμα που έχει ως στόχο να καλύψει τα πολύ δύσκολα εκκρεμώντα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν σε μια περιοχή που εξέρχεται από την σύγκρουση, από τη σύραξη. Αυτός ο πίνακας σας δείχνει την τάξη μεγέθους ε, και το εύρος των προγραμμάτων. Το PIS2 από μόνο του ε, είχε πάνω από 868.000 συμμετέχοντες και δραστηριότητες και πάνω από 161.000 από αυτούς συμμετείχαν σε διασυνοριακές πρωτοβουλίες. Αν γνωρίζετε τη Βόρεια Ιρλανδία, αν ξέρετε την ιστορία της Βορείου Ιρλανδίας, αυτά τα στοιχεία αυτά αυτά, είναι σημαντικότατα όσον αφορά την κλίμακα και τον αριθμό εκείνων που συμμετείχαν σε αυτού τις δραστηριότητε. Και αυτό δεν θα ήταν δυνατόν αν ευθύ παρεμβάσεω των προγραμμάτων PIS που επέφεραν σημαντική όθηση, πρόθεση και συνέβαλαν πάρα πολύ στην δευτική διαδικασία επιτόπου για πολλές δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Βοήθησαν επίσης τον κόσμο να ξανατοποθετηθούν, να αποφεληθούν από τις οικονομικές ε, δυνατότητες που ε, δημιουργούνταν στην περιοχή που ε, άρχισε να μπαίνει στην περιοχή της ειρήνης. Πού βρισκόμαστε τώρα στον αφορά το πρόγραμμα PIS 3 Έχουμε ένα πρόγραμμα που έχει τέσσερις πυλώνες. Ο πρώτος από αυτούς εστιάζεται στις κοινο... διάφορες τοπικές κοινότητες και πάνω από ένα τρίτο από το πρόγραμμα ασχολείται με αυτό το θέμα. Θέλουμε να έχουμε σε επαφή με τους τοπικά εκλεγμένους ερετούς εκπροσώπους των κοινοτήτων εκεί που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη πολιετών σχεδίων, για κοινοτικό σχεδιασμό, για την καλή ζωή των κοινοτήτων τους και για να δημιουργήσουν θετικές σχέσεις μεταξύ των κοινοτήτων σε πάρα πολύ τοπικό επίπεδο και αυτό ήταν επιτυχέστατο όσον αφορά αυτό το πρόγραμμα. Η τοπική αυτοδιοίκηση ε, συνεργάζεται σε συνολικό επίπεδο σε διάφορες ομαδοποιημένες προσπάθειες ε, διαπολιτικά, σε διακομματικό επίπεδο. Ο δεύτερος πυλώνας ασχολείται με τα θύματα και τις οικογένειες αυτών και τους επιζήσαντες της περίοδου των συγκρούσεων και πάρα πολλά αυτά τα χρήματα πάνε προς την παροχή βοηθείας αυτών των ανθρώπων. Τρίτος πυλώνας είναι πρακτική παρέμβαση με προγράμματα που δημιουργούν κεφάλαιο, ε, ώστε να δημιουργούνται κοινοί ε, δημόσιοι χώροι σε περιοχές οι οποίες ήταν απογορευμένες παλιά, όπου ήταν ανασφαλείς για τον κόσμο και θέλουμε να δημιουργήσουμε νέους κοινούς δημόσιους χώρους. Και ο τέταρτος πυλώνας είναι η δημιουργία δυναμικού για ένα κοινό μέλλον και πολύ συγκεκριμένα σε αυτόν τον πυλώνα του παρόντος προγράμματος έχουμε σαν στόχο να γίνει ανταλλαγή εμπειριών με άλλε περιοχές τη Ευρώπη διότι τώρα έχουμε σημαντική εμπειρία στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε έρθει σε επαφή με, με περιοχές όπως είναι η χώρα των Βάσκων, με την Κύπρο, επέδειξαν ενδιαφέρον τα Βαλκάνια, οι χώρες της Βαλτικής και είμαστε σε επαφή με διάφορα, διάφορες φορείς ειρηνευτικού στην Ευρώπη που θέλουν να μάθουν από τις εμπειρίες των προγραμμάτων PIS θέλουν να δουν πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αυτόν, πώς αυτό το μοντέλο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες ε, περιοχές. Βλέποντας πιο πρακτικά τα επιτεύγματα των προγραμμάτων PIS από το 2007 μέχρι τώρα, βλέπουμε ότι εξακολουθούμε τη διαδικασία ε, επαφών με τον κόσμο επιτόπου, με πάρα πολλούς συμμετέχοντες. Είμαστε ασχολούμαστε με πολύ δύσκολα και περίπλοκα ζητήματα δια, δια, ε, διασχιστικών τάσεων και ρατσισμού που ήταν πάρα πολύ δύσκολα προβλήματα για μας και τις επιτόπιες κοινότητες. Θέλαμε να αντιμετωπίσουμε τις διασυνοριακές δυνατότητες που δημιουργούνται και να ασχοληθούμε και με τις ανάγκες εκείνων που απαιτούν βοήθεια, αρρωγή ε, σε οικογενειακό επίπεδο, με τους συγγενείς τους για να αντιμετωπίσουν τα, διά, τα διάφορες τραυματικές εμπειρίες και μόνο τώρα ίσως να μπορούν να μιλήσουν για κάποιες από τις εμπειρίες τους και να προβάλλουν τις εμπειρίες τους και να ασχοληθούν με τις εμπειρίες τους. Ήθελα να σας δώσω, αν είχα επιλογή θα ήθελα να φέρω μαζί μου κάποιους εκπροσώπους των διαφόρων επιτοπίων προγραμμάτων, αυτό δεν ήταν δυνατόν, διότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θα ήθελα να σας δώσω μια γεύση των ε, θεμάτων με τα οποία ασχολούμαστε. Βλέπετε αυτή τη διαφάνεια, βλέπετε μια φωτογραφία ενός μεγάλου υψηλού τείχους, είναι ένας από, τους, από τα μεγάλα ψηλά τείχη που υπάρχουν ακόμα στο Belfast και σε πολλές κοινότητες στην Βόρεια Ιρλανδία λέγονται στίχοι της ειρήνης. Πολύ συχνά έχουν γραφίτι, έχουν ζωγραφιές, εικόνες πάνω τους και μπορούν να είναι πολύ προκλητικές. Τα τελευταία χρόνια ε, κάναμε πολλές προσπάθειες εργασία με τις κοινότητες και από τις δύο πλευρές των τυχών αυτών για να δημιουργήσουμε ένα πνεύμα εμπιστοσύνη ε, να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και σιγά σιγά σταδιακά να κατεδαφιστούν αυτή η τύχη, η φυσική αυτή τύχη και η ψυχολογική τύχη και η μεταφορική τύχη που εξακολουθούν να υπάρχουν και εξακολουθούν να είναι πολύ ισχυροί. Έχουμε ε, κάνει πάρα πολλή δουλειά με τους νέους. Αυτή η διαφάνεια εδώ δείχνει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που αφορά ε, ανθρώπους που είναι από 5 μέχρι 25 ετών και τους προσφέρουμε συμβουλές, στήριξη ψυχολογική και τους βοηθούμε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν κληρονομήσει λόγω των εμπειριών τους στην περιοχή να αντιμετωπίσουν την κληρονομιά των συγκρούσεων και βεβαίως αυτοί οι νέοι άνθρωποι είναι η μεγαλύτερη πρόκλησή μας για το μέλλον. Και εφόσον μιλούμε τώρα για το μέλλον, πιστεύω ότι με τους νέους θα πρέπει ε, να καταβάλουμε πολλές προσπάθειες για να αντιμετωπίσουμε τις ειδικές τους ιδιαίτερες ανάγκες. Αυτή τη διαφάνεια σας δείχνω μια φωτογραφία μιας γέφυρας μια γέφυρα που κατασκευάστηκε με τη βοήθεια του προγράμματος, διασχίζει έναν ποταμό στο Derry, London Derry και συνδέει δύο τμήματα της πόλης, τα οποία ήταν διαχωρισμένα αρχικά, όχι μόνο λόγω μέσω του ποταμού, αλλά από μακρά ιστορία, κουλτούρα, παραδόσεις. Είναι μια γέφυρα που φέρνει μαζί τις δύο πλευρές της πόλης και φέρνει το κέντρο της πόλης με, με διάφορα παλιά κτίρια που ήταν ε, καταβλισμός στρατιωτικός και ήταν Βρετανικός στρατός πριν, στο Derry, στο London Derry. Και εδώ να, είναι γέφυρα για πεζούς και ποδήλατα. Επίσημα θα εγκαινιαστεί αυτό το Σάββατο στις 25 Ιουνίου. Αλλά είναι πολύ ισχυρό σύμβολο, ισχυρή εικόνα των επιτευγμάτων, των προγραμμάτων της ειρήνευσης, πεις σε αυτό το μέσο του κόσμου και πολύ καλό παράδειγμα ε, των όσων έχουμε πετύχει. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα διαφόρων προγραμμάτων που σχετίζονται με τον αθλητισμό. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τι οικογένειε να ξανασυμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσει για να καταπολεμήσουμε το ρατσισμό και τα διάφορα απομονωτικά κινήματα μέσω αθλητικών εκδηλώσεων. Ε, συνεργαζόμαστε με τον κόσμο στις διάφορες ε, στις διάφορες γατικές κατοικίες. Εδώ έχουμε ένα πρόγραμμα που προσπαθεί να ενθαρρύνει ε, ολοκλήρωση, ένταξη στη στέγαση. Αναφέρθηκα στα τείχη ε, που χώριζαν τις κοινότητές μας και είχαμε κοινότητες που ήταν περιστοιχισμένες από τείχη και για να ρίξουμε τους φραγμούς και ενθαρρύνουμε τον κόσμο να έχει εμπιστοσύνη και να μπορεί να ζήσει με τους άλλους ε, πρέπει να καταβάλουμε πολύ σημαντικές προσπάθειες επιτόπου με αυτούς τους ανθρώπους και αυτή η δουλειά γίνεται ε, και είναι αποτέλεσμα, εφαρμόζεται χάρη στα χρήματα που διατίθεται μέσω των προγραμμάτων PIS. E ε, αυτά είναι παραδείγματα αυτών που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Αν δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον, εγώ θα σας έλεγα ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει, ε, δεν μπορεί κανείς να να ξεριζώσει τα βαθιά ριζωμένα προβλήματα τέτοιων συγκρούσεων που ζήσαμε στην Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία ε, μέσω δύο συντόμων προγραμματικών περιόδων, διορθώσαμε τις γέφυρες, ανοικοδομήσαμε τις πόλεις, ανοίξαμε τα σύνορα, αλλά οι καρδιές και τα πνεύματα του λαού, του κόσμου και οι σχέσεις μεταξύ των κοινοτήτων είναι ακόμα ένα σύνορο, είναι μια πρόκληση που είναι μπροστά μας. Ακούγοντα τα νέα από τη Βόρεια Ελλανδία χτε το βράδυ, αν είχατε ακούσει, θα βλέπατε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στι επαφέ μεταξύ των κοινοτήτων, σημεία διαπαφή. Θα ακούσατε διάφορε αποσχιστικέ ομάδε παραστατικές ομάδες που εξακολουθούν να αποτελούν ε, απειλή ε, επιτόπου. Άρα χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά και νομίζω ότι θα δείτε τα δύο κράτη-μέλη, η Βρετανία και η Ιρλανδία, δέχονται ότι, ότι υπάρχει ακόμα δυνατότητα να εξακολουθήσουμε αυτή την προσπάθεια στα πλαίσια του προγράμματος Peace. Το ειρηνευτικό αυτό πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίζει να εργάζεται με τις κοινότητες, να δημιουργεί εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινοτήτων, το, PIS, το, πρόγραμμα, το πρόγραμμα PIS θα πρέπει να καλύπτει τι ιδιαίτερες ανάγκε των νέων, εκεί επί τόπου, και να δούμε τι δυνατότητε που να δημιουργηθούν για αυτού, τι υπάρχουν. Πρέπει να στραφεί προ το μέλλον αυτό το πρόγραμμα, να δει τι δυνατότητε ε, έχουμε και αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο τώρα που βγαίνουμε από την ύφεση και υπάρχει μια έντονη χρηματοστική κρίση που πραγματικά έπληξε ε, την εμπιστοσύνη πολλών εκεί. Και νομίζω ότι θα θέλαμε ένα ε, πρόγραμμα ειρήνης που θα θα ήθελε συμμετοχή σε τοπικό επίπεδο και σε διεθνέ επίπεδο και προσβλέπουμε σε μελλοντικό πρόγραμμα να μπορέσουμε να μοιραστούμε, να συνεχίσουμε να ανταλλάσσουμε εμπειρίε με άλλου, ίσω με πιο δομημένο, διαθρωμένο, βαθύτερο τρόπο, να συνεργαστούμε με άλλε περιοχέ τη Ευρώπη. Εδώ έχω υπόψη μου ιδιαίτερα τα Βαλκάνια, τα νέα κράτη-μέλη, περιοχέ που εξακολουθούν να εμπεριέχουν πολλέ διαφορέ και μπορούν να δουν στην Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία τη δυνατότητα που υπάρχει να ωφεληθεί κανεί από τα διευθυντικά ταμεία, να τα κάνει να εργαστούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο που καλύπτει την κληρονομιά του παρελθόντο, τα προβλήματα, τι δυσκολίε. Ε, που απέρεσαν με τέτοια σύγκρουση όπω αυτή. Ευχαριστώ για τον χρόνο σα. ευχαριστώ εκ μέρου όλων τη Βορείου Ιρλανδία. ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη τη οποία τη είχαμε επί σειρά ετών μέσω αυτών των προγραμμάτων και προσβλέπουμε στη συνέχεια συνεργασία μαζί σα στο μέλλον επ' αυτών των θεμάτων. Σα ευχαριστώ. Thank you very much indeed. Ευχαριστούμε πολύ, Πατ. Θα περάσουμε αμέσω στον Τένι Ευρυνή. Εκτό μικροφώνου. Uh, σα ευχαριστώ. Προφανώς ε, βοηθήκαμε σε μεγάλο βαθμό από την Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της ε, Επιτροπής για το έργο που ανέλαβαν για μας. Ε, ιδιαίτερα προς το Ταμείο, το ενδιαφέρον των διαφόρων Ευρωβουλευτών ε, προ το Ταμείο μας. Σήμερα το απόγευμα θα ήθελα να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να αναφερθώ σε τρεις πτυχές του έργου του Ταμείου. Πρώτον, ε, το ιστορικό, δεύτερον κάποια κοινά σημεία της στρατηγικής και κάποιες σκέψεις για το μέλλον. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τους στόχους. Σύμφωνα με τη συμφωνία του 1986 ιδρύθηκε το Διεθνές Αυτοταμείο, ε, μια μοναδική οργάνωση. Έχει βεβαίως ε, ένα διοικητικό συμβούλιο και από τις ε, δύο μεριές ε, των συνόρων. Έχουμε πέντε διεθνείς δωρητές, όμως ε, η μεγαλύτερη συνεισφορά γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. στόχος, οι στόχοι του Ταμείου είναι εδώ πέρα μπροστά σας στην οθόνη να προωθήσει και την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και την ειρήνη όμως και τη συμφιλίωση και έχουμε πετύχει πολλά σε αυτόν τον τομέα. Το 2005 όμως αναγνωρίσαμε την ανάγκη να προσαρμοστούμε στις αλλαγές ε, ε, που υπάρχουν μετά την κατάπαυση του πυρός. Βεβαίως και την βελτίωση των οικονομικών συνθήκων και στις δύο πλευρές των συνόρων. και μέσω της στρατηγικής που καθορίσαμε εξακολουθήσαμε να αναπτύσσουμε πρωτοπόρες ε, στρατηγικές ε, σε διαφόρους τομείς όπως την παιδεία και το καθεξής για την δημιουργία βιώσιμων ε, δυνατήτων για ένα μοιρασμένο, ένα κοινό μέλλον. Θα συνεχίσουν αυτές οι δράσεις βεβαίως να έχουν θετικές επιδράσεις και μετά την λήξη του προγραμματός μας. έχουμε έρθει σε επαφή και με άλλε ζώνε συγκρούσεων, ιδιαίτερα στο ιστορικό της ε, Ευρώπης και ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία αυτή. Θα ήθελα να βρεθώ σε τρία, προγράμματα, ε, σε τρία παραδείγματα των ε, τρέχοντων δράσεών μας. Πρώτον, έχουμε την, δράση, την εκπαίδευση όπου υπάρχει διαχωρισμός σε επίπεδο 90% στη Βόρεια Ιρλανδία. Εμείς προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει εκπαίδευση σε, αυτόν, σε αυτή την περιοχή. Πρώτη δράση ήταν το πρόγραμμα ε, σεβασμούς προς τη διαφορά ε, που αφορούσε 5.000 παιδιά σε προσχολική ηλικία και 340 καθηγητές προσχολικής ε, ηλικίας ε, για να τους βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να, να τους αποστείλουμε μάλλον τα σωστά μηνύματα. Μετά χρησιμοποιήσαμε τα ειδικά σχολεία σαν ένα καταλήτη για την συμμετοχή σε αυτή την συζήτηση ιδιαίτερα επιτυχής ε, δράση και έχουμε ήδη φτάσει στα 60 σχολεία για τους 100 δασκάλους και 2.500 μαθητές. Αυτό και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα ε, πραγματικά έχουν επιφέρει τεράστιες αλλαγές ε, στην οτροπία του κόσμου. Συνεχίζω τώρα στις πρωτοβουλίες για την νεολαία. Το Ταμείο μας ε, έχει αναλάβει τέτοιες δράσεις από την αρχή της ύπαρξής του. Το πρόγραμμα το οποίο θα σας αναφέρω είναι το πρόγραμμα LET, Learning and Educating Together, και αφορά μαθητές 12-13 ε, ετών και από τις δύο ε, πλευρές των συνόρων, και από το βορρά και από το νότο. Το κύριο πρόγραμμα αφορά μαθητές 14 έως 16 ετών, ε, όπου οι μαθητές πηγαίνουν σε κατασκηνώσεις αλλά και μαθήματα ε, μετά το σχολείο, ε, όπου ουσιαστικά τους διδάσκουμε τη συμφιλίωση. Πέρσι υπήρχαν 900 νέοι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα και έτσι το θεωρούμε πρόγραμμα ιδιαίτερα επιτυχές. Το, δεύτερο, το τρίτο πρόγραμμα έχει να κάνει με το εξή. Υπήρχε τεράστια απόλωση στη στέγαση στην ε, Ιρλανδία μετά τις ε, σειράξεις ε, και έτσι δημιουργήθηκαν περιοχές με μία και μόνο ταυτότητα. Εμείς θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να αγκαλιάσουν αυτή τη διαφορετικότητα μέσα στην κοινωνία και έτσι να αυξήσουμε την κοινωνική ένταξη. Ε, αυτό ήταν πολύ θετικό γιατί οι ίδιοι πολίτες μπορούν να αποφασίσουν ε, το μέλλον τους αλλά σε διάφορες ε, πόλεις με 60.000 σε 60.000 κατοίκους πλέον αποδέχονται αυτό το πρόγραμμα και θα συνεχίσουμε και με περαιτέρω βεβαίως. Δεν έχω πολύ χρόνο να δώσω πολλά παραδείγματα, όμως αναφέρθηκα σε αυτά τα προγράμματα που έχουμε αναλάβει με ιδιαίτερη επιτυχία και αυτό αναφέρεται και σε πρόσφατη ανεξάρτητη αξιολόγηση και βεβαίως κάποιος θα συνεχίσει ε, αυτό το έργο. Θα φτάσουμε στα, τώρα φτάνουμε στα μελλοντικά μας ε, σχέδια. Υποβάλαμε μία ε, τελική έκθεση το 2008 Ε, όπου αναφέρουμε και τα προγράμματα που θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Τα τελευταία χρόνια βεβαίως και η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν θερμιολαιόδου σημασία στην επίτευξη των στόχων μας, όμως ακόμα μένουν πολλά να γίνουν. Ε, κάθε μέρα βλέπουμε παραδείγματα που μας επενθυμίζουν ε, την πόλωση που υπάρχει και τον διαχωρισμό που υπάρχει ανάμεσα στις κοινότητές μας. Υπάρχουν κοινότητε που ακόμα δεν έχουν επιφεληθεί τη της ειρηνευτική διαδικασία. Ε, το 2010 το Ταμείο ε, προσέλαβε έναν εξωτερικό σύμβουλο ε, για να συστήσει ένα καινούριο πρόγραμμα για να βοηθήσει αυτές τις ιδιαίτερες περιοχές που ακόμα δεν έχουν επιφεληθεί των αλλαγών. Έχουμε εντοπίσει τέσσερις κύριες περιοχές. Θα σας δώσω μια μικρή γεύση αναφερόμενος σε μία περιοχή, που, ε, το Λέργαν, 30 λεπτά από το ε, Belfast, με 30.000 κατοίκους. Ε, πριν από τις Ιράξεις, οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες ζούσαν δίπλα-δίπλα, όμως μετά την σύγκρουση είχαμε τεράστιες αλλαγές. Βλέπετε και στις διαφάνειες τις διαφορές που υπάρχουν πλέον από το 1970 μέχρι σήμερα. Υπάρχει συνεχής ε, δράση παραστατικών οργανώσεων και ε, συνεχή βία γεγονότα. Οι εικόνες που βλέπετε εδώ πέρα ήταν από πέρσι. Επομένω, ο σύμβουλος ε, τον οποίο προσλάβαμε δείχνει ότι υπάρχουν πάρα, πάρα πολλά προβλήματα σε αυτές τις περιοχές. Κάτι που μπορεί να μας βάλει μέσα σε έναν αρνητικό ή και καταστροφικό κύκλο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη αυτή την ερνητική διαδικασία να αναφερθώ ε, σύντομα σε αυτή τη, στα προβλήματα. Ε, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, ανεργία, χαμηλό επίπεδο ανασχόλησης, ε, ε, εντάσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες και βία. Ε, ε πόλωση, ρατσισμός, περιθωριοποίηση των νέων απώλεια ή μάλλον έλλειψη υποδομών για τους νέους, εγκληματική δραστηριότητα, βεβαίως ε, απόσταση από ε, την ειρηνευτική διαδικασία και αποδοκιμασία της ε, κυβέρνησης και του πολιτικού κόσμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να φτάσουμε σε αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές ή μάλλον στις ε, δυσπρόσιτες περιοχές και με την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει μέχρι τώρα μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν γέφυρα και να συνδέσουμε τους, ε, ε, τους διαφόρους φορείς ε, της κοινωνίας. Ε, πάντα να έχουμε έναν ηγετικό ρόλο σε αυτό το τομέα και να διασφαλίσουμε ότι οι πόροι που μας δίνονται δεν κατανέμονται με πολιτικά κριτήρια. Ε, βεβαίως έχουμε και τη στήριξη και της Ιρλανδικής και της Βρετανικής κυβέρνησης, αλλά και των δύο κοινοτήτων. Θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω προγράμματα, τρία στη Βόρεια στην Ιρλανδία και άλλο ένα στην, ε, στην Ιρλανδία. Εμείς θα προτείνουμε νέες οργανώσεις και νέες ε, διευθυντικές ομάδες που θα αντιμετωπίσουν αυτά τα ενδυμικά προβλήματα. Πάντα σε στενή συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Για μας αυτό είναι το τελικό τμήμα της λειτουργίας μας, αλλά χωρίς περαιτέρω χρηματοδότηση ε, θα μείνουν ανολοκλήρωτα αυτά τα προγράμματα. Εμείς είμαστε πιστός συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πολλά χρόνια. Ε, και ω τέτοιο έμπιστος εταίρος σας συμβουλεύουμε γιατί εμείς έχουμε πολύ ε, σημαντικό έργο ακόμα να επιτελέσουμε για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Commission. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στην ε, Επιτροπή, στην Διευθυντή Αντρές. Παρακαλώ να είστε όσο το πιο σύντομος, γιατί Έχουμε πολλές συζητήσεις ακόμα. Πείτε μας μόνο τα πιο σημαντικά σημεία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας. Πράγματι είναι υπερήφανη, πολύ υπερήφανη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμμετέχει ενεργά σε αυτές τις πρωτοβουλίες με καλά αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Και είχαμε συμμετοχή επί 22 έτη στο ΑΙΦΑ και αντίστοιχα μεγάλη θητεία στο πρόγραμμα Peace, Ειρήνη. Βρισκόμαστε στη διαδικασία του να κλείσουμε το ΆΙΦΑ αυτή τη στιγμή. ΆΙΦΑ ε, έχει καταδείξει ένα πραγματικά πολύ ικανό επίπεδο δράσεων, πολύ κοντά στις κοινότητες όπως προαναφέρθηκε από τον Ντένις. Δίνει πολύ καλά αποτελέσματα αυτά και η μεγάλη επίπτωση στην καθημερινή ζωή είναι σε σχέση με τους ίδιους τους πολίτες, συνεισφέροντας για την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης, επενδύοντας τους νέους, εξυγχρονίζοντας τις υποδομές ε, και τον εξοπλισμό, δημιουργώντας τη βάση για την αηφορία στην ανάπτυξη. Ένα καλό παράδειγμα είναι αυτό το παράδειγμα για αυτή τη γέφυρα που θα ε, εγγενιαστεί ε, σύντομα και δυνατότητα να είναι παρόντες σε άλλα μέρη της Ευρώπης και να συμμερίζονται τα βιώματά τους και πολύ σημαντικό αυτό και για το άμεσο μέλλον. Τέλος, Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω κάτι, το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ καλά συνειδητοποιήσει ότι η διαδικασία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχουν πουλωθεί οι πληγές και υπάρχουν πολλές φορές εκρήξεις βίων πράξεων, βιοπραγιών βλέπουμε ότι υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει ακόμα για να εμπεδοθεί η ειρήνη και η συμφιλίωση. Και πραγματικά είμαστε ευγνώμονες για τις τεράστιες προσπάθειες μέχρι σήμερα όλων των εμπλεκόμενων που συνεισέφεραν στη σαφή επιτυχία της ειρήνης και της διαδικασίας συμφιλίωσης. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Ανοίγει ο γύρος τώρα για τις παρεμβάσεις. James Nicholson, παρακαλώ. Thank Uh, Ευχαριστώ. Δεν το άνεμενα ότι θα ήμουν ο πρώτος. Αφού είσαστε ο πρώτος πρέπει να είσαστε πολύ σύντομος γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Ελπίζω να μην είσαστε πολύ αυστηροί μαζί μου πρόεδρε γιατί έχω αρκετά πράγματα που θα ήθελα να πω. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές που, που συνεισέφεραν με τις παρεμβάσεις τους για την συνεισφορά τους με τον κύριο Ρούνη δεν είχα τόσες ε, πολλές επαφές, αλλά με τον Πατ, ο Πατ και εγώ είχαμε πολλές συναντήσεις ε, και επαφές. Κάποιες από αυτές ε, συμφωνούσαμε, κάποιες άλλες διαφωνούσαμε. Θέλω να αποτίσω φόρο τιμή στην εξαιρετική δουλειά που ο Πατ και οι συνάδελφοί του έκαναν αυτά τα χρόνια και κάτω από δυσχερέστατες συνθήκες και σε δύσκολη συγκυρία. Δεν θα επαναλάβω τίποτα από αυτά που προαναφέρθηκαν. Σίγουρα πρέπει να πω ότι η Βόρεια Ιρλανδία έχει καλύψει πολύ μεγάλη απόσταση από εκείνα τα παλιά χρόνια για το IFI όταν ξεκίνησε και το Peace Funds όταν ξεκίνησε και θυμάμαι και πάντα θα το λέω όταν ξεκίνησε αυτό από κοινού με τον John Hume, τον Wesley και εμένα είμαστε τα άτομα που προσπαθούσαν τότε να κάνουν κάτι και ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια των ετών. Τούτων λεχθέντων η Βόρεια Ιρλανδία όμως εξακολουθεί να είναι ε, επίκεντρο για τα όσα συμβαίνουν και τα γεγονότα, τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να μας κάνουν να οπισθοχωρήσουμε, να γυρίσει ο χρόνος πίσω. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να επιστρέψει η Βόρεια Ιρλανδία στην περίοδο του ζόφου τη σκοτεινή εκείνη περίοδο. Πρέπει να πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της Βόρειας Ιρλανδίας δεν θέλουν να οπισθοδρομήσουν. Θέλουν να προοδεύσουν, θέλουν να κινηθούν προς τα εμπρός, δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν στο παρελθόν με, αυτές, με αυτόν τον τρόπο που κάποιοι επιθυμούν. Θέλω να πω κάθετα και ξεκάθαρα ότι η ιστορία του PIS 1, PIS 2 και PIS 3 είναι ποικίλη υπήρξαν πολλές καλές δράσεις ε, και για το ποιος έκανε τι υπάρχουν ίσως ε, κάποιες διαφωνίες και όταν ε, έχουμε λιγότερα κονδύλια είναι δύσκολο να υπάρξουν και πολλές νέες προτεραιότητες. Δεν είναι, πολύ, δεν είναι καθόλου εύκολο να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Όμως οι συνάδελφοι και φίλοι στην Ευρώπη μου είπαν επανειλημμένα και το ξέρουμε αυτό ότι πόσο καιρό χρειάζεται για να επιτευχθεί η ειρήνευση. Και πάντα λέω ότι υπάρχει αυτή, αυτό το θέμα και πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες. Θέτω αυτό το θέμα σε σχέση με τον Πατ Κάουντον και το κατέστησε σαφές ε, ο κύριος ε, Ρούνε ότι το ΑΕΦΑ θα ε, ολοκληρωθεί αλλά θα υπάρξει παράταση ή επέκταση του peace, της προσπάθειας αυτής πέρα, από αυτό το στενό πλαίσιο γιατί είναι κάτι που πρέπει να αξιολογηθεί σωστά και να ε, εξεταστεί αυτή η προοπτική και σίγουρα βρίσκεστε υποπίεση χρόνου και δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο πρόεδρε θα θέλω όμως να σας πω ότι έδωσε αξία και πρόσθετη, ε, έδωσε κέρδη και ωφέλη και υπήρξαν περίοδοι, πολλές περίοδοι όπου δεν μπορούσε κανείς να αξιολογήσει ποια ήταν ε, αυτά τα ωφέλη. Αυτή είναι η διαφορά αυτών που κάνουμε και το, του έργου που στο, στο οποίο εμπλεκόμαστε εμείς. Ένα τμήμα μιας ολόκληρης διαδικασίας που εξελίσσεται και πρέπει να εξελιχθεί, μια και είχε τέτοια προϊστορία, πρέπει να τύχει συνέχεια. Ξαφνικά βλέπουμε, για παράδειγμα, κάποιους που λένε έχω χρήματα σε σχέση με το ε, Peace Fund δεν ήξερα αυτό σχετικό, ούτε θα ήξερα αν αυτό το επιχείρημα ευσταθεί ή όχι. Πρόσφατα στο IFA που είχα πάει στο Belfast μου είπαν για τη δουλειά που κάνουν εκεί και το τι γίνεται για την αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων σε σχέση με ποδοσφαιρικές αθλητικές συναντήσεις. Εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει εκεί και τι φόρο τιμής σε αυτούς που συμμετείχαν σε αυτό το έργο και όλους όσους εμπλεκόντουσαν σε σχέση με το παρελθόν υπήρξε κάποια ανησυχία όταν είπα κάποια πράγματα στο παρελθόν. Εγώ πιστεύω ότι ως πολιτικός δουλειά μου είναι να διατυπώνω δύσκολα ερωτήματα πέρα από το υπόλοιπο έργο μου. Θα ήθελα να ε, πω στους εταίρους ότι η ειρήνη και η συμφιλίωση δίνει σήμερα ίδια αποτελέσματα όπως στο παρελθόν. Ξέρουμε ότι ε, ο σχεδιασμός που είχε γίνει στο παρελθόν μεταξελίχθηκε. Πολλά έχουν γίνει και προχώρησαν και τι φόρο τιμή σε αυτά. Ξέρω ότι πραγματικά στο αξίωμά σα πρόεδρε η... Πάντα προσπαθώ να σέβομαι τον, πρόεδρο, τον προεδρεύοντα ή την προεδρεύουσα, αλλά είναι ένα θέμα που πρέπει να γνωρίζετε ότι έχει τεράστια σημασία για μας και αν πρέπει να συνεχιστεί θα πρέπει να έχει την υποστήριξη υποχρεωτικά και την εμπιστοσύνη και των δύο κοινοτήτων και σίγουρα έκανε πολλά στη διασυνοριακή πτυχή. Συμφιλίως έφερε κοντά ανθρώπους που ποτέ δεν θα είχαν προσεγγίσει ο ένας τον άλλο. Με αυτό το πνεύμα προσεγγίζω και ευχαριστώ για αυτό το έργο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ότι θα, θα είσαστε και εσείς υπόδειγμα για τους επόμενους ομιλητές. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την δυνατότητα που δίνετε να μιλήσω σήμερα. Όπως οι δύο μιλητές από τη Βόρεια Ιρλανδία είπαν, η Βόρεια Ιρλανδία προχώρησε πάρα πολύ. Είναι ένα καλύτερο μέρος τώρα από ό,τι ήταν πριν από 10-20 χρόνια. Και το Ταμείο αυτό για την Ειρήνη έδωσε προστιθέμενη αξία. Δεν ήταν τέλειο, αλλά έχει προστιθέμενη αξία και συνέβαλε σημαντικά στην προσέγγιση των κοινοτήτων και οι κοινότητε αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες. Παραμένουν όμως ακόμα προβλήματα στη Βόρεια Ιρλανδία και δημοσία ε, η ομάδα ιστορικών ερευνών στη Βόρεια Ιρλανδία που συνδέεται με τι αστυνομικέ υπηρεσίες της Βόρειας Ιρλανδίας θα υποβάλει έκθεση όσον αφορά τη σφαγή στο Kings Mill. Σφαγιάστηκαν άνθρωποι εδώ και κάποια χρόνια. Εργα εργάτες, ε, τους τραβήξαν από ένα λεωφοριάκι και τους εξετέλεσαν. Ε, στο County Down στη Βόρεια Ιρλανδία, στο Lohan Island, θα δοθούν τα πορίσματα μιας έρευνας σχετικά με τι έγινε με τους δικούς τους συγγενείς όταν βασιλόφρονες ε, μπήκανε σε μια πάμπα και πυροβόλησαν αθώους. Παραμένουν πάρα πολλές δυσκολίες και είχαμε διάφορες ε, δραστηριότητες. Πυροβολήθηκαν δύο στρατιώτες ε, πριν φύγουν για το Αφγανιστάν. Ο Στίβεν Κάρολ και ο Ρόμαν Κέιρ ε, πυροβολήθηκαν. Και ο, ο Πρωθυπουργό Κάμερον ήρθε στη Βόρεια Ιρλανδία την περασμένη εβδομάδα και είπε ότι από το 2006 κάτι που δεν αναγνωρίζεται εύκολα. Το 2006 ο αριθμός από 37-48 αποθήματα. Ακόμα και σε περίοδο σταθερότητας οι κοινότητες βρίσκουν δυσκολίες να ζουν δίπλα ημέν στους δε και ψώνουν τύχη. Ε, αν θέλουμε να δούμε τι έγινε στην, ε, τι έκαναν τα προγράμματα ποιης, e πρέπει να το δούμε αυτό, αλλά πρέπει να δούμε πώς να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα των προγραμμάτων ποιης για να επενδύσουμε για το μέλλον. Προσέξτε και μία περιοχή του Belfast που εκπροσωπούσε επί σειρά ετών. Την περιοχή Σάνκλ. Κυρίως προτεστάντες είναι εκεί. Εάν στεκόμαστε αυτόν τον δρόμο, 70% από όλες, από όλες φόνους στη Βόρεια Ιρλανδία έγιναν σε μια κτίνα 2 μιλίων από εκεί που θα στεκόμουν. Έχει βαθιές ρίζες το πρόβλημα σε αυτές τις κοινότητες υποφέρουν από χαμηλή εκπαίδευση, ε, υψηλή ανεργία, κακή υγεία και εδώ θα πρέπει να επενδυθούν χρήματα του ΠΙΣ για το μέλλον, να επενδυθούν χρήματα για τους νέους. Και αυτό ταιριάζει και με τους στόχους του 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να το υπερασπιστούμε σαν στόχο. Πρέπει να συμμετάσχουν οι νέοι μέσω κατάρτισης, παιδείας, δυνατοτήτων να βρουν δουλειά, Πρέπει να δούμε και οι γυναίκες τι ρόλο που απέξουν στην Βόρεια Ιρλανδία. Οι γυναίκες μπορούμε διατομιακά να εκπαιδεύσουμε τις γυναίκες και να τις καταρτήσουμε. Σε μελλοντικές συζητήσεις για το ΠΙΣ, πρέπει να δούμε ποιοι έχουν υποτιμησιακή πρόσβαση στη χρηματοδότηση να επαναξεταστεί αυτό. Ομάδες ε, πρώην φυλακισμένων, Φερρυπίν. Το 1994 έγινε η πρώτη κατάπαυση του πυρός. Το 1998, σε συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, απελευθερώθησαν οι κρατούμενοι. Και πρέπει να διατηρηθεί η Ευρώπη πότε κανεί σταματά να είναι πρώην φυλακισμένος και πότε ξεκινά να είναι πολίτης. Σημαντικότατα ζητήματα αυτά πρέπει να ληφθούν οι υπόψη στην αξιολόγηση των πεπραγμένων και προσβλέποντα προ το μέλλον. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ, Σον Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αρχικά πρέπει να πω ότι θετικό ήταν που ο συνάδελφο Νίκολσον αναγκάστηκε να μιλήσει σήμερα, γιατί συμμετείχε και με τον John Hume και τον Dr. Pierce εκείνη την πρωτοβουλία. Βεβαίως ως ηγητής για το Κοινοβούλιο αναγνώρισα τα ωφέλη και είχα ε, την τιμή πριν από μερικούς ε, μήνες να συζητήσω με τον συνάδελφο Εγώ πολλές φορές, πολύ συχνά πηγαίνω στην ε, Βόρεια Ιρλανδία, ενώ ένας άλλος ε, μέχρι πρόσφατα δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό να πάω σε συγκεκριμένε περιοχές εκεί. Και μάλιστα με υποδέχτηκαν και θερμά. Και ήταν πολύ καλό αυτό που είδα εκεί, δηλαδή αυτή την, ε, αυτές, την επαφή που υπάρχει πλέον μεταξύ των κοινοτήτων τοπικά σχολεία και ούτε καθεξής. Και ότι αυτό συνεχίζεται πέρα από το IFR και το πρόγραμμα Peace. Η ειρήνη βεβαίως δεν είναι διασφαλισμένη και μάλιστα μόλις χθε υπήρξαν ε, ορισμένες ε, ε, αναταραχές στον Παλιφάστ. Το θέμα εδώ είναι ότι απαιτείται συνέχιση για το PIS4. Και όπως είπε και ο Ντένις Πατ, στις ε, δυσπρόσθετες περιοχές όπου, που αποτελούν ε, γόνιμο έδαφος για, τους, ε, για αυτές τις αποσχιστικές ομάδες. Ενδεχομένως, αν συνεχίσουμε με ένα πρόγραμμα PIS4, να απομακρυνθούμε από αυτούς τους κινδύνους. Ε, Πρόσφατα είχαμε και την προσωπία των ΗΠΑ που υπογράμμισαν την, ε, την ε, δράση του IFR σε αυτό το τομέα και εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε αυτή την χρηματοδότηση. Και βεβαίως όλα τα μέρη θα θέλουν να συνεχιστεί αυτή τη διαδικασία. Γιατί ταιριάζει απόλυτα και με τη στρατηγική για το 2020, αλλά και με τις αρχές που είχαν καθορίσει οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Σούμαν και οι υπόλοιποι. Έτσι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Τέλος, ήθελα να πω ότι σήμερα το πρωί που συνάντησα τους συναδέλφους, ανέφεραν και τον ρόλο που διαδραματίσετε εσείς, Πρόεδρε, σε αυτή τη διαδικασία, οπότε σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πατ Γκάλαγκερ, τέλος. Uh, Καταρχάς, Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στο έτοιμά σα να συντηθείτε με εκπροσώπου του, του Φορέα για τα Ειδικά Προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ενώση και το IFI. Ευχαριστώ εκείνου που συνέβαλαν, τον Μπατ Κόριγκαν και τον Ντένι Ρίλε. Η σημερινή συνεδρίαση με φέρνει πίσω στο 2001 όταν είχαμε συνεδριάσει εδώ όταν πρώην πρόεδρος του IFI και ο Πάτι Χάρτ που είναι εδώ σήμερα ήρθαν προσπαθώντας να πείσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα έπρεπε να συνεχίσουν την παροχή χρημάτων. Έγιναν και εκθέσεις. Ο Higgins το 2006 θα έκανε μία. Τι θυμόμαστε τις εκθέσεις αυτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητήθηκε να εγκρίνει χρηματοδότηση προς τη Βόρεια Ιρλανδία και παραμεθόριες κομιτείες, είτε μέσω του IFI ή του PIS. E δεν υπήρχε κανένας βουλευτής που να ήταν αντίθετος και κανείς δεν είχε απόσχει τότε. Αυτό είναι προς τιμήν της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το 1985-86 είχε συναυθεί συμφωνία. Ποιο έπαιξε σημαντική, σημαντικό ρόλο τότε. πρώην Πρωθυπουργό Ελλανδία, που πέθανε πρόσφατα, ο Γκάρεθ Φιτζέραλτ, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτή τη συμφωνία. Και ευχαριστούμε και τον Ζακ Δελόρ. διότι την παραμονή της πάσης των εχθροπραξιών ο Ζακ Δελόρ αμέσως αν, αντέδρασε και είπε ότι θα τη δράσει η Ευρώπη θετικά. Θα μπορούσαν να είναι απλώς λόγια, αλλά αμέσως. Αύξησε την εισφορά προς το Εθνικό Ταμείο για την Ιρλανδία και δημιουργήθηκε ε, η προσπάθεια συμφιλίωσης. Ε, ήμουνα με τον Jim Nicholson, τον Dr. Paisley και τον John Hume σε ένα γεύμα τότε που δημιουργήθηκε αυτή η προσπάθεια. Το IFI και το PIS διαφέρουν. Προσπαθούν όμως να πετύχουν τον ίδιο στόχο. Ε, διαφέρουν πολύ. Το Wi-Fi ήταν κάτι πιο απτό. Το PIS προσπαθούσε να συμφιλιώσει κόσμο, όπως έλεγε και ο Πατ Κόριγκον. 41.000 μόνιμες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν και έμεσες 70.000 απασχόλησης δημιουργήθηκαν τότε. Συνεχίζεται αυτό, ίσως όχι στην διακλίμακα. Δεν θέλω να χρονοτριβήσω. Θέλω να πω πόσο σημαντικό είναι να συνεχιστούν και το PIS, και το 4 και το Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία επί σειρά Θεωρείται γιατί πρέπει να συνεχίσουν οι ΗΠΑ να δίνουν χρήματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγραψε σε πολλού φίλου τη Ιρλανδία, στο Κογκρέσο και στη Γερουσία και ζήτησαν την υποστήριξή του να δώσουν και άλλα χρήματα. Αν δώσουν του πόρου οι Αμερικανοί, θα δίνουν και άλλοι πόροι. Εάν δεν δώσουν αυτοί τα χρήματα, αυτό δεν είναι δικαιολογία για την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση ή για την Ιρλανδική κυβέρνηση, την Βρετανική κυβέρνηση να μην, να μην δώσουν. Πρέπει να συνεχιστούν τα προγράμματα. Εγώ ανατριχιάζω όταν σκέφτομαι τι θα χρειαζόταν να χρειαστούμε νέα νομοθεσία. Δεν πρέπει να αλλάξουμε νομοθεσία επί σειρά ετών. Μπορούμε να το κάνουμε βάσει της παρούσης νομοθεσίας να συνεχίσουμε να αναθεωρηθεί. Ενθουσιάζομαι από την ιδέα της ανταλλαγής εμπειριών με άλλε χώρε. Αναφέρθηκε η χώρα των Βάσκων, η Κύπρο, τα Βαλκάνια και άλλε χώρε. Στη Βόρεια Αφρική μπορούμε να μοιραστούμε εμπειρίε μαζί του. Δεν χρειάζεται να επανεφευρεθεί ο τροχό. Έχει εφευρεθεί στη Βόρεια Ιρλανδία mm. και στι ε, παραμεθόριες έχουν και οι δύο κυβερνήσεις, ο Πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο μας, έχουν υποβάλει αίτηση για συμπροματικούς πόρους για να προχωρήσουν τα προγράμματα. Είναι ερώτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντική η σημερινή συνεδρίαση. Πρέπει πιο τακτικά ίσως να επαναλαμβάνεται αυτό και να γίνονται και πιο τακτικά επισκέψεις στις Βρυξέλλες, να έρχονται εκπροσωποί της Ιρλανδίας, <coughs> όπως είδαμε και στις διαφάνειες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα να συναντώμαστε και με τι ομάδε που ωφελούνται από μας. Εγώ με τον Τόνε Γκόλ από την άλλη μεριά των συνόρων. Ατλαντικό από τη μία, Βόρεια Ιρλανδία από την άλλη. Δεν υποφέραμε στον ίδιο βαθμό βέβαια όπω η Βόρεια Ιρλανδία από πλευρά ανθρώπινη, Οικονομικά όμω, έχουμε υποφέρει. Διότι όποιο έρχεται από την υπόλοιπη χώρα ταξιδεύει από τη Βόρεια Ιρλανδία. Και εγώ είμαι υπερήφανο εκπρόσωπο περιοχή και εκπρόσωπο των μια κομιτεία από την αλυσίδα των κομιτιών που είναι παραμεθόριος για τη δουλειά που έγινε για την ε, ε, ειρήνευση. Εμεί ω εγωιστέ πολιτικοί θέλουμε να εξακολουθήσει η χρηματοδότηση και το ΑΕΦΑΙ και το ΠΙΣ να συνεχίσουν την καλή τους δουλειά και ενδεχομένω να είναι πιο εστιασμένη η προσπάθεια, να είναι ε, πιο σαφεί οι που θέτονται από τα προγράμματα. Πολύ σύντομα, Πατ. Ε, Σε ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα αν επιτρέπετε να πω κάτι. Η πρόοδος που επετέφθη ως αποτέλεσμα των προγραμμάτων για την ειρήνη μπορώ να αναλώσω μεγάλο χρόνο αναφέροντας, αλλά δύο παραδείγματα να δώσω. Την εμπλοκή των ερετών εκπροσώπων στις τοπικές αρχές στην Βόρεια Ιρλανδία και στις ε, μεθοριακές ε, κομιτείες έχουν διοργανωθεί σε οκτώ ομάδες, οκτώ ομάδες ε, τοπικών αρχών που συντάσσουν, καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα δράσεων για τις σχέσεις μεταξύ των κοινοτήτων. Το ίδιο γίνεται και σε σχέση και με τις κομιτείες ε, κατά μήκο των συνόρων. Αυτό δεν θα μπορούσε να είχε γίνει χωρίς ε, το πρόγραμμα για την ειρήνη. Τεράστια πρόοδος έχει επιτευχθεί. Δεύτερο παράδειγμα. Τόσες πολλές πόρτες άνοιξαν, που ήταν κλειστέ επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και τόσο πολλοί, τόσοι πολλοί άνθρωποι συνομιλούν μεταξύ του που στο παρελθόν δεν ήταν δυνατόν να έχουν επαφέ Και όταν υπάρχουν ταραχε, υπάρχουν άτομα και από τι δύο κοινότητε, πέρα από τη γραμμή, την, τη διαχωριστική γραμμή που κατεβαίνουν στον δρόμο και προσπαθούν να υποπτεύσουν και να αστυνομέσουν ώστε να είναι ήρεμο ε, το κλίμα. Και αυτό είναι κάτι μοναδικό και είναι κάτι που αξίζει να διασφαλιστεί για το μέλλον. Και να πω, αναφέρθηκε επίσης τι θα εμπεριέχεται σε ένα νέο πρόγραμμα για την ειρήνη. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι δεν υπάρχουν κάποιες προκατηλημένες απόψεις και ιδέες ιδεολειπτικά. Μια ευρεία διαδικασία διαβούλευσης θα απαιτεί για να συμπεριληφθούν οι ανησυχίες και να καλυφθούν αυτά τα οποία αναφέρθηκαν από τους προλαλήσαντες και να ληφθούν υπόψη τα μελήματα αυτών που ζουν κατά μήκος των συνόρων. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του μελλοντικού προγράμματο για την ειρήνη θα είναι, όπως είπαμε πιο πριν, τα κοινά αυτά βιώματα που πρέπει να επεκταθούν σε ευρύτερη βάση. Α ολοκληρώσω προσκαλώντα τα μέλη τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή, όταν το θεωρήσετε σκόπιμο, να έρθετε να μα επισκεφτείτε ξανά στη Βόρεια Ιρλανδία, όπω το κάνατε και στο παρελθόν. Και να έρθετε να δείτε πώ είναι οι δρόμοι μα, ποιο είναι το κλίμα εκεί και να δείτε τι υπάρχει και τι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ξέρω ότι κάποιοι το κάνατε στο παρελθόν. Θα καλωσορίζαμε ιδιαίτερα μια νέα επίσκεψη στι οδού του Μπέλφαστα και στην υπόλοιπη Βόρεια Ιρλανδία για να δείτε οι ίδιοι από πρώτο χέρι με τα μάτια σα ότι έχει σημειωθεί πρόοδο αλλά υπάρχει και μεγάλο έργο που πρέπει να καλυφθεί. Σα ευχαριστώ. Εσεί θα θέλετε να πείτε δύο λόγια για να ολοκληρώσετε. Παρακαλώ. Απλά να πω πρόεδρε ότι πιστεύω ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να απαντήσουμε το ερώτημα είναι μια περίπτωση να ζητάμε περισσότερα κονδύλια απλά επειδή μπορεί να πάρουμε κάποια χρήματα ή να τονίσουμε ότι εμείς δώσαμε δώσαμε πολύ φροντίδα και σκέψη σε αυτό το θέμα ως ζήτημα. Πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αναλώσαμε να δούμε τι πρέπει να γίνει για αυτά που είναι σημαντικά για μας και με τη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους στις κοινότητές μας για όλα αυτά και μετά από αυτές τις διαβουλεύσεις δεν θα είχαμε επιστρέψει σε εσά εκτός αν πιστεύαμε ότι αυτή η διαδικασία ήταν σημαντικό να συνεχιστεί αυτό το σημαντικό έργο δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή, διαβουλευτήκαμε με όλους τους εμπλεκόμενους και αφού αποφασίσαμε και διαβουλευτήκαμε για αυτούς τους λόγους καταλήξαμε στο ότι είναι σημαντικό για μας να απευθύνουμε αυτή την έκκληση να συνεχιστεί η υποστήριξη για το έργο που επιτέχθηκε στο παρελθόν και πρέπει να συνεχιστεί. Ε. Σα ευχαριστούμε. Να ενημερώσω του συναδέλφου που ήρθαν με καθυστέρηση ότι αυτή η ακρόαση για του ε, δύο αρμόδιους για την υλοποίηση των προγραμμάτων για τη Βόρεια Ιρλανδία που είναι το πρόγραμμα για την ειρήνευση Peace Program μέσα στο πλαίσιο τη περιφερειακή πολιτική Κόλγαν ε, και Ρούνι από την Διεθνή Πρωτοβουλία για την Ιρλανδία όπου και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη συνεισέφεραν τα τελευταία χρόνια και είχαμε αυτή την ακρόαση επειδή θα λάβουμε σοβαρές αποφάσεις μετά τις θερινές διακοπές για το μελλοντικό πλαίσιο αυτής της πολιτικής για την διαπεριφερειακή συνεργασία, όπου έχουμε φιλοδοξίες ως επιτροπή, ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή και για την αύξηση κονδυλίων και ζητήσαμε να δούμε, να έχουμε πληροφορίες για το πώς αυτά τα προγράμματα, ποιες επιπτώσεις είχαν και τι επέτυχαν και πρώτα απ' όλα πώ βλέπετε εσείς ίδιοι την ανάγκη να συνεχιστούν αυτά τα δύο προγράμματα στο μέλλον. Αυτές οι πληροφορίες είχαν τεράστια σημασία, ήταν σπουδαιότατε. Ελπίζω θα είμαστε σε επαφή και ελπίζω ότι αυτή η πρόσκληση, αυτά τα στοιχεία που υποβλήθηκαν θα ληφθούν όλα υπόψη στις διαβουλεύσεις μα ε, κατά το επόμενο διάστημα, στα χρόνια που έχουμε μπροστά μας είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα αυτά στη δράση μας και πρέπει να τα λάβουν οπωσδήποτε υπόψη. Και πάλι σας ευχαριστούμε που προσήλθατε στο Ευρωκοινοβούλιο. And Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της σημερινής τη διάταξης, στις ψηφοφορίες. Σήμερα το πρωί δεν ε, το ελέγξαμε. Πρέπει να δούμε λοιπόν αν ε, λειτουργούν τα μηχανήματα. I'm so far. I'm here. Okay, can we open? Uh, We are voting already. Okay. Αρχίζει η ψηφοφορία λοιπόν. Ελέγχουμε τα μηχανήματα. Yeah. Δεν μπορούμε να κλειδώσουμε την ψηφοφορία γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των ψηφισάντων και του αριθμού που βλέπουμε εδώ. Ξεκινάμε λοιπόν ε, με την ε, έκθεση στα βρακάκι. Είχαμε 41 τροπολογίες και έχουμε καταλήξει και σε ένα σύνολο συμβασμών. Ξεκινάμε λοιπόν την διαδικασία για την τροπολογία αριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Συμβασμός 1. Υπέρ. Κατά. Και πάλι. Συμβασμός 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. Συμβασμό 6 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. Συμβασμό 2 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. Περνάμε στο συμβασμό 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. Συμβασμός 9. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμός 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμό 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμό 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμό 8. 8 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Συμβασμός 9, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Περνάμε στην τροπολογία 23, υπέρ, κατά, αποχές, Ε, Τροπολογία 24, υπέρ, κατά, Ελέγχουμε για την τροπολογία 24, ένταξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Τροπολογία 26, υπέρ. Κατά. Αποχές, υιοθετείτε. 28, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Συμβασμός 10, υπέρ κατά, αποχές, υιοθετείτε. Τροπολογία 30, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε, 31 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε, 33 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 38 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Και μετά τελική ψήφος ηλεκτρονικά, άνοιξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. 36, 4 αποχές. Χαρητήρια. So now we go to... This one, okay, sure. So uh, Ψηφίσουμε τώρα την ε, γνωμοδότηση Olbricht. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, ελέγχουμε. Δεν ξέρω αν υιοθετήθηκε. Ε, Έναξη ψηφοφορίας. Πέρας. Υιοθετείτε. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 11. Υπέρ. Κατά. Ε, για να ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται νομίζω. Ας ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Με 29 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμός 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16. 60, 18. Υπέρ. Τροπολογία 18. Α, 16 μου λένε... Α, τον απορρίψαμε. 16 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 18 τώρα λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές Υιοθετείτε. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 2 υπέρ κατά αποχές Υιοθετείτε. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές Υιοθετείτε. 24 Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 31 υπέρ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, δεν ξέρουμε. Ας ελέγξουμε. Τροπολογία 8. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Τροπολογία 38 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε επί της ψηφοφορίας ηλεκτρονικά. Επί της ονοματότητας, συγγνώμη. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Συγχαρητήρια. Ολοκληρώνονται πέρα ψηφοφορίες. Ας περάσουμε στην ακρόαση τώρα. Είναι όλοι παρόντες ή η Επιτροπή δεν έχει φτάσει ακόμα. Συνάδελφοι, θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτό το χρονικό διάστημα για να ανακοινώσω τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τους συντονιστέ σήμερα το απόγευμα για την ε, κατανομή γνωμοδοτήσεων και εκθέσεων. Οι σοσιαλιστές θα ελέγξουν αν ε, τους ενδιαφέρει να αναλάβουν τη γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ε, Ε, για τις Κανάριες νήσους. Εάν όχι, τότε θα το αναλάβει η Προεδρία. Δεύτερον, για τον οδικό χάρτη για μια νέα ευρωπαϊκή ε, ε, περιοχή μεταφορών πάει στους σοσιαλδημοκρατές. Ε, κανόνες γενικού οικονομικού συμφέροντος θα ελέγξει η Προεδρία αν ε, αφορά αυτό την ε, δική μας επιτροπή και αν ναι θα το αναλάβει η Προεδρία γιατί οι ομάδες δεν έχουν αναλάβει, ε, δεν έχουν δείξει ενδιαφέρον. Για το gender mainstreaming, Elizabeth Schroeder πρότεινε η Προεδρία να, να υπογράψει επιστολή με την γνώμη της Επιτροπής Reggie μετά για το νομοθετικό πλαίσιο για την συνοχή μετά, πολιτική συνοχή μετά το 2013 έχουμε λάβει τις εξής αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά τον γενικό κανονισμό δεν έχουμε ακόμα τελική απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων. Παρ' όλα αυτά αποφασίσαμε ε, να έχουμε ε, σοσιαλδημοκράτες και Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σαν ε, εισηγητές. Εάν ε, η απόφαση είναι αρνητική, τότε θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα. Για τον κανονισμό και το EDF πήγε στο ΕΛΚ για το Ταμείο Συνοχή του Σοσιαλιστέ, για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Συνεργασία στο Άλντε, για το EGDC στο ΕΛΚ, για την γνωμοδότηση για τα κοινωνικά ταμεία Πάμε ε, στους σοσιαλδημοκράτες. Για το πολιετές ε, ε, πλαίσιο η γνωμοδότηση θα προετοιμαστεί από το ΕΛΚ και για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο δεν ξέρουμε ακόμα τη νομική διαδικασία που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ECR εξέφρασαν ενδιαφέρον, αλλά ακόμα δεν μπορούσαμε να πάρουμε απόφαση. Μετά συζητήσαμε το ζήτημα της έκθεσης πρωτοβουλίας Ιδία πρωτοβουλία, Δύο ε, αποφασίστηκαν. Μία πρόταση ΕΛΚ, τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις ε, εξωτερικές περιοχές στο πλαίσιο της ε, θετικής 2020 και μετά ο ρόλος των δημοσίων προμηθειών στην πολιτική συνοχή. Οι σοσιαλιστές εκδήλωσαν ενδιαφέρον να παρουσιάσουν σύντομα μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας και επίσης το ΕΛΚ πρότεινε το 2000 να υποβάλουν έκθεση ε, εφαρμογή για το 2011 για την αναθεώρηση της στρατηγικής για την Βαλτική. Για τις εξωτερικές ε, μελέτες ε, μένει ανοιχτό το θέμα. Προς το παρόν έχουμε έξι συνεχιζόμενες εκθέσεις και τον Ιούλιο ελπίζουμε να προτείνουμε μία νέα καινούρια εξωτερική, εξωτερική μελέτη Προς το πάνω θα το χειριστεί η Γραμματεία και η Πολιτική Συμβουλή και μετά θα δούμε τι θα αποφασίσουμε τον Ιούλιο. Ας κλείσω εδώ λοιπόν τα νομιωτικά. Είναι εδώ όλοι ενδιαφερόμενοι για την εξωευρωπαϊκή διάσταση. Η Επιτροπή επικυρώνει τα, τις αποφάσεις των συντονιστών. Λάμπερτ, συμφωνεί. Εντάξει. Επομένω, συμπεραίνω ότι η Επιτροπή υιοθετεί τις αποφάσεις των συντονιστών. Προς το παρόν περιμένουμε τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συζητήσουμε αυτές τις τρεις ε, εκθέσεις. που προετοίμασε. Να περάσουμε σε κάτι άλλο. Α, η κυρία Σμολκοβάιτς. Οι σκιώδες είναι εδώ. Uh, Ο κύριος Ουσπάσκης δεν είναι εδώ, δεν ξέρουμε αν θα έρθει. Οι σκιώδες δεν έχουν έρθει. Ίσως να μην έρθουν και αργότερα βέβαια, αλλά...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 Να μην χάσουμε όμως ε, χρόνο έτσι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με το πιο σημαντικό από όλα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 23 εκατομμύρια ανέργους στην Ευρώπη και αυτό σε σχέση με τις ε, νέες θέσεις απασχόλησης είναι τεράστια σημασία ώστε η στρατηγική του 2020 να μπορέσει να υλοποιηθεί για την απασχόληση λαμβάνοντας υπόψη ε, τους από τους πέντε στόχους τρεις ε, είναι μετρήσιμοι και αφορούν και την κατάρτιση, εκπαίδευση και την απασχόληση στην οποία στοχεύουν. Και μάλιστα όχι τρεις αλλά τέσσερις από τους πέντε. Θα ήθελα να τονίσω ότι η έκθεση της κυρίας Μπάστος πρώτα απ' όλα ήταν πολύ επικοδομητική και με πολύ καλή ε, δουλειά που έγινε έχει διατυπωθεί. Τη δική μου γνωμοδότηση ήδη γραπτός την έχω καταθέσει, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, όμως ως πρώην δασκάλα ή καθηγήτρια θα ήθελα να τονίσω ότι η εκπαίδευση και η παιδεία είναι έχει τεράστια σημασία όσον αφορά όλες τις βαθμίδες, όσον αφορά την διαβίου μάθηση και εκπαίδευση και κυρίως την δέσμευση σε σχέση με τις σημερινές ανάγκες που πρέπει να προσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Δεν έχει αρκετά προσοντούχους εργαζόμενους η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τέτοιους προσοντούχους εργαζόμενους. Ωστόσο όμως πρέπει να γνωρίζουμε και να έχουμε συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν και μη προσοντούχοι εργαζόμενοι και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν για αντικειμενικούς και υποκειμενικούς λόγους. Και ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΡΕΓΙ για την περιφερειακή πολιτική και την ανάπτυξη, θέλω να στρέψουμε το βλέμμα στο γεγονός ότι τα κονδύλια, τα δημοσιονομικά μέσα πρέπει να χρησιμοποιούνται το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, ώστε να ακολουθούμε νέες δυνατότητες και δράσεις για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τα ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο για την διαβίου μάθηση και εκπαίδευση, για την επιμόρφωση και κατάρτιση των εργαζομένων, ώστε και στις μικρές επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι να μπορούν να προσαρμόζονται και να προετοιμάζονται. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να συμμετέχουν και στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο. Πρέπει όλα αυτά τα ταμεία να επικεντρώσουν τις ε, δράσεις τους στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Πιστεύω ότι η κατάρτιση, η εκπαίδευση, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης είναι δράσεις, είναι μέτρα που απαιτούν νέα κονδύλια. Αυτά τα κονδύλια πρέπει από κοινού να δρουν και να συντονίζονται όχι μόνο από τα ευρωπαϊκά ταμεία αλλά και ιδιωτικά κεφάλαια πρέπει να συστρατευτούν και να ενεργοποιηθούν ώστε να βαίνουν εκ παραλίλου στις προσπάθειες αυτές. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα ποσοστά απασχόλησης στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Γι' αυτό είναι αναγκαίο όλα τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν και να προαγάγουν αυτό το πρόγραμμα, ώστε τα θετικά βιώματα, η θετική πείρα που συλλέξαμε κατά το παρελθόν, έχουμε θετικές εμπειρίες και από τη Γερμανία και από την Αυστρία, όσον αφορά την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, όσον αφορά ιδιαίτερα τους νέους, που αποκτούν νέες δεξιότητες για να προσαρμοστούν στις ανάγκες ε, των, αγορών, όλα αυτά πρέπει να προαχθούν. Έχετε λοιπόν γραπτό στην γνωμοδότησή μου συνάδελφοι, προσβλέπω και χαίρομαι για τις παρατηρήσεις που θα κάνετε και τα σχόλια. Uh, e Ευχαριστώ για το ΕΛΚ, Γιώσεφ Ματούλα, πρώτος Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η γνωμοδότηση έχει τεράστια σπουδαιότητα θα έλεγα. Και τώρα θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποιες λίγες πτυχές των θεμάτων αυτών. Πρώτον, πρέπει να πω ότι πρέπει οπωσδήποτε να αεξεύρουμε την αναγκαία ισορροπία μεταξύ κατάρτισης και εκπαίδευσης αφενός, διότι μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μεριμνούμε για τη σωστή προετοιμασία και προπαρασκευή των εργαζομένων. Ισορροπία λοιπόν στη χρήση κονδυλίων από τα γνωστά ευρωπαϊκά ταμεία Πρώτα απ' όλα τοποθετούμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το ε, ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης. Όλα αυτά πρέπει να εξετάζονται από κοινού με το πρόγραμμα Progress και από κοινού με το πρόγραμμα διαβίου μάθησης και εκπαίδευσης, επιμόρφωσης. Ταυτόχρονα πρέπει και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να τύχουν της αναγκαίας προσοχής από πλευράς μας, διότι εφόσον δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης δημιουργούνται στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει υποχρεωτικά αυτός ο τομέας να τονωθεί να ενδυναμωθεί από εμά. Χαιρετίζω την ατζέντα, την ημερήσια διάταξη για τι νέε δεξιότητε και προσόντα ω τμήμα, ω μέρο τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Και αν θέλουμε να μεριμνήσουμε για μια αηφορία στην ανάπτυξη και καινοτομία για την ανάπτυξη, χρειαζόμαστε προσοντούχου, καλά προετοιμασμένου και εκπαιδευμένου εργαζόμενου ω εργατικό δυναμικό. Ακόμα πρέπει να δούμε και το θέμα της υπεργύρασης της ευρωπαϊκής κοινωνίας και να μην αγνοήσουμε τις δημογραφικές αυτές εξελίξεις όσον αφορά τη συρρήκνωση του πληθυσμού και τα θέματα μετανάστευσης. Αυτά με οδηγούν εν τέλει στην παρατήρηση ότι πρέπει να βρούμε την ισορροπία που χρειάζεται μεταξύ της άρσης των νομικών και τεχνικών προσκομμάτων και εμποδίων ώστε να φροντίσουμε ώστε να δημιουργηθούν επαρκείς θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί όχι να υπάρξει μια μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και των ε, προσόντων και πτυχίων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί. Θέλω να ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία στην εκπόνηση της νομοδότησης. Σπάνσκι για την δεν θέλετε να μιλήσετε. Η κυρία Ουκατσιεύσκα έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Σμόλκοβα για αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή. Θα ήθελα να φέρω ένα θέμα το οποίο δεν συμπεριελήφθη στην έκθεση και θα έπρεπε να έχει συμπεριληφθεί. Λόγω της ε, υψηλής ανεργίας που επικρατεί ανάμεσα στους νέους και τους προσοντούχους. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το τονίσουμε, καθώς θα πρέπει να τονίσουμε και τις ίσες ευκαιρίες ε, για τις γυναίκες στην αγορά εργασίας, διότι είναι σε μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας και οι γυναίκες. Οι Πρόεδρος, ε, δεν έχουμε άλλον που θέλει να πάρει το λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πει κάτι. Όχι, τίποτα. Λαμπέρ Φων Λίστερροι να πω μια σκέψη. Σημαντική. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε τον ανταγωνισμό, να γίνει ανταγωνιστική η Ευρώπη, να αναφερόμαστε στην παιδεία. Ε, το σχολείο και παιδεία είναι το κλειδί. Πρέπει να πούμε πιθανόν δύο πράγματα. Αυτό που βλέπω στη χώρα μου, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, βλέπω ότι υπάρχει ένα εθνικό πρόγραμμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι να έχουμε αποκεντρωμένη, ολοκληρωμένη εφαρμογή. Είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει σχέση μεταξύ με το Περιφερειακό Ταμείο και το Κοινωνικό Ταμείο. Και αν υπάρχουν δύο εντελώς διαφορετικά υπουργεία, όπως τη Γερμανία που υπάρχει αυτός διαχωρισμός, μεταξύ υπουργείων. Εάν είναι διαχωρισμένα τα υπουργεία δεν λειτουργεί το σύστημα είναι ε, ε, τόσα πολλά χρήματα. Ε, έπρεπε να υπάρχει μια πιο συντονισμένη προσέγγιση. Να το κάνουμε αποκεντρωμένα, σε κοινό πλαίσιο και να το ζητήσουμε. Και έχουμε και την έκθεση της κυρίας Βέσφαλ. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για τις ικανότητες εκείνων που είναι πιο μεγάλη από 50-55. Δεν είναι μόνο θέμα εργασίας είναι θέμα νοοτροπίας να παραμείνουν στη δουλειά. Ε, να κρατάνε ισορροπία εργασίας και άλλων μεταξύ εργασίας και άλλων δραστηριοτήτων που έχουν μεγάλη σημασία. Πολλοί στην Ευρώπη σταματάνε ή το θέλουν ή όχι να δουλεύουν στα 55. Και οι νέοι στόχοι είναι πολύ ψηλοί. Έχουμε τη γύρανση του πληθυσμού. Πρέπει να είναι συγκεκριμένο στόχος. Όλοι οι νέοι πρέπει να δουλέψουν. Και αν δείτε στατιστικές θα δουλέψουν. Χρειαζόμαστε όλα τα χέρια, χρειαζόμαστε όλα τα μυαλά την επόμενη 20 αιτία. Βλέποντας τις δημογραφικές αλλαγές. Τεράστιος στόχο θα είναι αυτοί που είναι περίπου που είναι στα 55 και πάνω και έχουν εταιρείε που έχουν συγκεκριμένη πολιτική γι' αυτό. Είναι καταστροφικό. Εξακολουθούν να, να ακολουθούν αυτή την τάση και να σταματήσουν την τάση. Η κυρία Βέσφαλερ έχει δύο, μία, δύο πολύ σοφέ τροπολογίε η ίδια. Δεν έχει πάρει το λόγο, είναι παρούσα, αλλά ίσω και εγώ μπορώ να κάνω κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Λαμπέρ. Κάποιο άλλο θέλει να μιλήσει. Η κυρία Σμόλκοβα, θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει πολύ λίγος χρόνος για την κατάθεση τροπολογιών θα είμαι όμως σε επαφή με τους σκιώδεις εισηγητές και χαίρομαι για την περαιτέρω συνεργασία μαζί τους. Ευχαριστώ. I Πολύ σημαντικό. Αυτό έχουμε πολύ σύντομα την προθεσμία υποβολή τροπολογιών, οπότε παρακαλώ τους σκιώδεις ηγητές και όλους τους συναδέλφους που θέλουν να εμπλουτίσουν την έκθεση και να επεκτείνουν την εμβέλειά τους μέχρι 22 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα λοιπόν τις τροπολογίες. Αύριο μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ελάχιστο χρόνο έχουμε για την υποβολή τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Σμολκόβα. Ολοκληρώνουμε αυτό το θέμα και μπορούμε να μπούμε στην ακρόαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διεθνής έξω ευρωπαϊκή διάσταση της περιφερειακής πολιτικής είναι το θέμα. Ας ακούσουμε πρώτα Ραφαέλ, τους Ραφαέλ Γκουλέ και Charles White. Μετά ακολουθεί ανταλλαγή απόψεων και αν έρθει και ο Πίτερ Μπέρκοβιτς θα ακούσουμε και την τρίτη παρουσίαση. Ραφαέλ Γκουλέ λοιπόν ξεκινάς. Uh, Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή που έχουμε να υποβάλουμε έκθεση σε εσά που είναι σωστό και δίκαιο σε σχέση με το έργο μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που οφείλεται στο τέλος τέλος στην υποστήριξη που παρέχεται από το Ευρωκοινοβούλιο επί δύο χρόνια, 2009 και 2010, μέσα στο πλαίσιο ενός ε, μιας ε, ε, προγραμματισμένης δράσης και τώρα μέσα στη, σε ξεχωριστή δράση. Προχωρούμε σε σχέση με τις εταιρική, την εταιρική συμφωνία και εταιρική σχέση με την Ρωσία, την Κίνα, τη Βραζιλία και συνεισφέρουμε και για την πρωτοβουλία σε σχέση με την γειτονική ανατολική σχέση με την Ουκρανία 2009 και πιο πρόσφατα με τη Μολδία τη Μολδαβία και τη Γεωργία. Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η επίσημη έναρξη του διαλόγου δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη συνεργασία μαζί μας, είναι μάλλον η επισημοποίηση και αναγνώριση της πολιτικής βούλησης που υπάρχει και είναι δεδομένη για την περιφερειακή πολιτική από κοινού και κάνοντας αυτό συνεισφέρουμε και στον ευδιάκριτο χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνει την ευκαιρία να μοιραστούμε διεθνώς την πείρα που έχουμε σε σχέση με την ε, οικονομική ανάπτυξη από πλευράς Ευρωπαϊκής ε, ε, Ένωσης. Μια δυνατότητα που δίνει την δυνατότητα να πούμε ότι βασιζόμαστε στις ανοιχτές αγορές στο σεβασμό του περιβάλλοντος, στην εφαρμογή των αρχών της πολιτικής για την ανάπτυξη και εδώ δεν κάνουμε λόγο μόνο για εμάς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το ευρωπαϊκό επίπεδο που συνεμπλέκεται κάνουμε λόγο και δείχνουμε ε, ανάγλυφα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές περιφέρειες ε, το έργο που επιτυγχάνεται. Δεν είναι τίποτα καινούριο, γνωρίζετε αυτά εσείς ήδη, πράγμα που δείχνει πολύ καλά το τι επιθυμούμε να κάνουμε, ε, θέτοντας ερωτήματα για την περιφερειακή πολιτική και σε σχέση με τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πώς μπορεί να γίνει όχι μόνο για τη Ρωσία, Ουκρανία και Κίνα αλλά επίσης μεταφράζεται και στα αρμενικά στα στην... για τη Γεωργία, την Αρμενία και αυτό δείχνει το πρόσφατο ενδιαφέρον αυτών των χωρών να εμπλακούν. Συνολικά σε όλα αυτά που κάνουμε προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την υποστήριξη αυτής της προκαταρκτικής ε, δράσης που μας δίνει όθηση επιπρόσθετα για να προχωρήσουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με όσα γινόντουσαν στο παρελθόν. Χάρη σε αυτή την υποστήριξη έχουμε τη δυνατότητα να παράσχουμε ένα ολόκληρο εύρος υπηρεσιών και δράσεων που δεν θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε διαφορετικά. <clears throat> Δεν είναι τίποτα εντυπωσιακό, αλλά αφορά την χρήση ε, διασκέψεων, συνεδρίων και από αυτό το πλαίσιο σε πιο επικεντρωμένες στοχοθετημένες δράσεις και χρησιμοποιώντας το μέσο των επισκέψεων μελέτης ή διαρευνητικών επισκέψεων σε σχέση με αυτές τις χώρες. Μια ιδιαίτερα αξιόλογη εμπειρία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάναμε 2009-2010 μέχρι σήμερα. Ξεκίνησε ο νέος διάλογος με την Μολδαβία και τη Γεωργία Συμφωνήσαμε προγράμματα δράσης με αυτές τις χώρες μέχρι σήμερα, όμως εδώ αντιμετωπίζουμε κάποιες, κάποια προβλήματα πολιτικής αστάθειας πρέπει να ομολογήσω και αλλαγές όσον αφορά τις πολιτικές δομές που σημαίνει ότι δεν βρισκόμαστε στο ύψος των φιλοδοξιών και των απαιτήσεων σε σχέση με αυτές τις χώρες. Ε, δεν είναι εύκολο να ε, καλυφθεί όλο αυτό το εύρος. Την επόμενη εβδομάδα θα πάμε στη Μολδαβία, θα έχουμε ένα σεμινάριο σε σχέση με ε, την εξέταση συγκεκριμένων χωρών και περιφερειών για να επεξηγήσουμε πώς λειτουργούν αυτές οι αρχές και πώς η περιφερειακή πολιτική δρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά το σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι η Ουκρανία όπου βλέπουμε αλλαγή υπουργού, ο Υπουργείου σε σχέση με την ε, περιφερειακή ανάπτυξη. Όχι, δεν είναι λόγο του διαλόγου μας που ξαφνικά αποφασίστηκε, να, ε, ε, αποφασίστηκε η κατάργηση του Υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο αναλαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Ελπίζουμε να έχουμε σύντομα επαφές με τους νέους υπεύθυνους για τις νέες δραστηριότητες ε, με τον ε, ΟΑΣΕ και με τις ε, δυνατότητες να συμμετάσχουμε στην Ουκρανία, να υπάρξει μια καλή επισκόπηση ποιες, ποια είναι τα πιο αδύνα, η πιο αδύναμη, αδύνατη κρίκη της αλυσίδας και ξεκινήσαμε το 2009 στις Βρυξέλλες με μια διάσκεψη και συνεχίσαμε μετά με δραστηριότητες για να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίηση. Ψάχνουμε να βρούμε στο συγκεκριμένους τρόπους για να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των εμπλεκόμενων χωρών, αιτήματα που έχουν διατυπωθεί και τα επιτυχή παραδείγματα που έχουμε είναι η συνεργασία με τη Βραζιλία μέχρι σήμερα όπου σίγουρα θεωρούμε ότι η συνεισφορά μας είχε επίπτωση στην προετοιμασία της δεύτερης πλέον φάσης της ε, βραζιλιανικής περιφερειακής πολιτικής και βλέπουμε αυξημένο αριθμό εμπλεκόμενων και από πλευρά των εταίρων μας σε σχέση με τα αρμόδια Υπουργεία και τη συμμετοχή διαφορετικών Υπουργείων αλλά και την συμμετοχή άλλων κρατικών εκπροσώπων όλα αυτά αντανακλώνται και σε σχέση με τον αριθμό των εμπλεκομένων αλλά και στα θέματα που εμπλέκονται. Πέρα από τα θέματα γενικής πολιτικής εξειδικευόμαστε και σε θέματα χειροπιαστής στοχοθετημένης πολιτικής. Πράγμα το οποίο εμπλέκει και το Βραζιλιάνικο Ελεγκτικό Συνέδριο. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς ε, σε σχέση με τις, ε, την λογιστική αυτές οι δραστηριότητες ταιριάζουν και με τις, ε, τα όσα γίνονται και σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό που προανέφερα, αν κάποιοι από εσάς δεν συμμετέχετε άμεσα στην ε, υλοποίηση κάποιων από αυτές τις δράσεις, πιστέψτε μας ε, ότι σε σχέση με τους ε, αρμοδίους αυτών των χωρών γνωρίζουν το τι συμβαίνει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτή η υποστήριξη πάντα αναφέρεται στις δράσεις που αναπτύσσουμε. Και αυτό αντανακλάται σίγουρα εξάλλου και στην πιο συνολική ανταλλαγή απόψεων στα πιο σφαιρικά ε, θέματα που εξετάζουμε στις επισκέψεις μας. Ποιες είναι οι προτεραιότητες. Προφανώς πολιτικά ε, φέτος και τα επόμενα έτη θέλουμε να θέσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ανατολική γειτονική σχέση και στην πολιτική γειτονία γενικά. Έχουμε αυτές τι επαφές με την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία όπως προανέφερα. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση θα θέλαμε να εμπλακούν και κάποιες από τις χώρες σε επίσκεψη αποστολή αυτή τη κοινοβουλευτική Επιτροπής με 20 Ουκρανούς εκπροσώπους που θα έρθουν να επισκεφθούν τέσσερις διαφορετικές χώρες εδώ σε μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεχίσουμε το έργο μας σε σχέση με την ανάπτυξη των ήδη θεσμοθετημένων διαλόγων με τη Βραζιλία, με την Κίνα επίσης. Θέλω να τονίσω αυτή τη νέα δράση που αναπτύσσουμε μαζί τους ένα μείγμα επισκέψεων μελέτης και διερευνητικών επισκέψεων που δίνουν ε, γενικές ε, την εικόνα των αρχών ε, και το, του πώς μπορούν να εφαρμόζονται αυτές οι πολιτικές. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη συμμετοχή του κυρίου Φανίστερ Ρόι σε αυτές ε, τις ε, δραστηριότητες ε, που έγιναν για πρώτη φορά τον Μάρτιο εφέτος και παρότι είναι δύσκολο σε αυτή τη φάση να κρίνει κανείς και να αξιολογήσει ποια θα είναι τα τελικά αποτελέσματα αυτού του διαλόγου είναι, σχετικά, είναι αρκετά ενδιαφέρον να δει κανείς ότι οι Κινέζοι σκέπτονται πώς θα είναι δυνατόν αυτή η ανάπτυξη να τύχει συνέχεια εμπνέονται σε σχέση με την προσπάθεια ε, περιοχών και σύγκλησης όπου υπάρχουν κοινά στοιχεία. Δεν θέλω εδώ να πω ότι αυτό είναι αποκλειστικό αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου, αλλά τέτοιου είδους συνεργασία και ανταλλαγές απόψεων επιτρέπουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα ή μια τέτοια εξέλιξη. Με τη Ρωσία στρατηγική σημασία σε τέρο, έχουμε μεγαλύτερες δυσκολίες στις επαφές. Ενώ θέλουμε να υπάρχουν αυτές οι επαφές οπωσδήποτε και θέλουμε να αποκομίσουμε το μέγιστο από αυτές τις επαφές. Έχουμε ένα πλέγμα μόνο το στο πω έτσι, ε, δραστηριοτήτων ή ε, αστικών κέντρων ή πόλεων ε, σε σχέση με τις πιο σχετικά πιο ενδιαφέρουσες ε, ευρωπαϊκές εμπειρίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης. Επακούμε σε αυτές τις παρατηρήσεις και προσβλέπω στις παρατηρήσεις τις δικές σας, στα σχόλιά σας και ερωτήσεις σας. Να δώσουμε το λόγο τώρα στον Τσάρλ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμπληρώσω ε, τα, στα όσα είπε ο Ραφαέλ. Η βοήθεια που λάβαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την ε, πολιτική ευρωπαϊκής ε, γειτονίας υπάρχουν εξελίξεις στα προγράμματα που περιλαμβάνουν προγράμματα, πιλωτικά προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης αλλά για να ξεκινήσει αυτός ο διάλογος ήταν θεμελιώδη σημασία ε, η συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων. Να φτάσουν δηλαδή να έρθουν αυτοί οι εμπειρογνώμονες στην Ευρώπη. Μόνο και μόνο για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Επομένω, ε, μα βοήθησε ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ανάπτυξη αυτών των στρατηγικών ε, πρωτοβουλειών. Και τώρα έχουμε στρέψει το βλέμμα όχι μόνο προ ε, την Ανατολή, αλλά και προ τον Νότο, για να δούμε μήπω μπορούμε να αναλάβουμε αυτέ τι δραστηριότητε και για την, για την Τινησία, το Μαρόκο, όπου έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την πολιτική. Έχουμε ήρθει, ήδη έρθει σε επαφή μαζί του και αυτό ήθελα μόνο να πω ότι ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη συνεισφορά του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Από ό,τι κατάλαβα, Πίτερ θα πάρει το λόγο αργότερα. Μπορούμε λοιπόν να δώσουμε τώρα στον Λάμπερτ Βανίστελ Ρόι. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι μια παράδοση, μια φορά το χρόνο, να συζητάμε για την ε, πρόοδο που σημειώνεται στα πιλωτικά σχέδια και τις δράσεις. Ε, αναφερθήκατε σε ένα έγγραφο, αλλά δεν το έχω εγώ στα χέρια μου. Ίσως να μην το έχω λάβει μόνο εγώ, ίσως να το έχετε εσείς, Πρόεδρε, δεν ξέρω. Θα βασιστώ στα όσα άκουσα. Το σημαντικό είναι να δούμε αν υπάρχουν απτά αποτελέσματα, συγκεκριμένα αποτελέσματα Αναφέρθηκατε σε μία επίσκεψη στην Κίνα στο πλαίσιο ενός προγράμματος ανταλλαγής. Πώς ε, θα χειριστούμε την πολιτική συνοχή, την πολιτική γυτνίασης, ε, αλληλεγγύης σε μια χώρα όπου υπάρχουν πολιτικη γυτνίαση, αλληλεγγυης σε μια πόλεις ε, με τεράστια ανάπτυξη και αστικοποίηση. Βλέπουμε λοιπόν εκεί τι έχει κάνει και η Ευρώπη ή τουλάχιστον το ενδιαφέρον που παρουσιάζεται να κοιτάξουμε τι έχει γίνει στην Ευρώπη. Το Λονδίνο για παράδειγμα, ε, μέσα στην ε, πολιτική αυτή ε, τονώνει και προωθεί άλλες οικονομίες ε, στην διαδικασία αυτή. Για παράδειγμα η Ευρώπη έχει γίνει πιο δυνατή, βοηθώντας και άλλες οικονομίες. Και αυτό είναι το μυστικό της Ευρώπης. Μεγάλη φιλοφρόνηση βέβαια αυτή όταν το ακούμε από άλλους. Έχουμε πλέον τόσα πολλά προγράμματα και, ε, και τόσα πλαίσια στήριξης και ανάπτυξης που βοηθούν και στην ανάπτυξη των ε, κινέζικων αστικών κέντρων. Αυτό θα ε, αναπτυχθεί περαιτέρω και στις, ε, σε αυτό το Open Days που θα γίνει στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο. Πολύ σημαντική εκδήλωση και αυτή. είναι κρίμα βέβαια γιατί το το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι να κοιτάξουμε μαζί με την Κίνα πώς ε, διεξάγουν αυτή την, την πολιτική cluster policy. Και μετά βεβαίως εκεί θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα επενδύσουν ε, και ο ΣΑ και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και στο τέλος της χρονιάς είδαμε ότι τελικά δεν έγινε κάτι, δεν έγινε αυτό το βήμα. Καταλάβαμε λοιπόν ότι ε, στην επιφάνεια υπάρχει βούληση, αλλά μόλις εμφανιστούν προβλήματα σταματάει. Θα ήθελα λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν να ακούσουμε κάτι παραπάνω από αυτού. η Κίνα και η Ινδία μας ρωτούν πώς ακριβώς ε, ακολουθούμε μια πολιτική των μεγάλων αστικών κέντρων και των Μητροπόλεων. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο παραπάνω γι' αυτό. Μετά τι συμβαίνει με τη χρηματοδότηση. Εμείς δίνουμε κάθε χρόνο ένα ποσό. και με βάση πρωτοβουλίας ε, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Λοιπόν, τι συμβαίνει με αυτό. Τι συμβαίνει με αυτή τη χρηματοδότηση. Ίσως βλέπουμε ότι ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουμε, ας πούμε, αντιμετωπίζουμε και με τη Ρωσία Εκεί πέρα λοιπόν θα πρέπει να, να υπάρξει μια αναπροσαρμογή στις προτεραιότητές μας. Όπου δηλαδή τα πράγματα πηγαίνουν, πηγαίνουν καλά, να δώσουμε με μεγαλύτερη έμφαση. Τι γίνεται λοιπόν με την κατανομή των πόρων. Και τέλος, ε, σας έστειλα και μια επιστολή, ε, ρωτώντας αν είστε διατεθειμένοι ε, να λάβετε υπόψη στο ίδιο επίπεδο τις ε, τη διεθνή διάσταση, την υπερευρωπαϊκή διάσταση και το καθεξής. Θα ήθελα να ξέρω αν μπορούμε όλα αυτά να τα δούμε πιο σφαιρικά. Θα ήθελα όμως ένα κείμενο για να τα έχω και μπροστά μου. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω για την παρέμβαση που έγινε από τους ε, πραγματογνώμονες σήμερα. Και να πω το εξής. Κανονικά κάθε φορά που κάνω παρεμβάσεις σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή σε σχέση με τις υπερπεριφερειακές ε, περιοχές παραδέχομαι ότι κουράζονται πολλές φορές οι συνάδελφοι γιατί είναι επαναληπτικές αυτές οι παρατηρήσεις για τις διαρκείς δυσκολίες και μόνιμες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υπερπεριφερειακές περιοχές. Όμως σε αυτή την περίπτωση πέρα από την το συσχετισμό σε αυτές τις δυσκολίες που είναι πραγματικές δυσκολίες και μόνιμες δυσκολίες, σήμερα πρέπει να κάνουμε λόγο για μια άλλη πρόπτικη που προσπάθησα να παρουσιάσω στη συζήτηση το ότι αυτές οι περιοχές δεν έχουν μόνο αυτούς τους περιορισμούς, αλλά έχουν και δυνατότητες και ένα μεγάλο δυναμικό. Και αυτό είναι ένα τέλειο παράδειγμα εδώ του δυναμικού που έχουν οι υπερπεριφερειακές περιοχές της Ευρώπης ότι βρίσκονται και εντοπίζονται σε ένα γεωγραφικό χώρο που πολλές φορές αμελούμε εμείς όλοι μας. Δηλαδή ιδιαίτερα όσον αφορά τη γειτονική σχέση τη γυτνίαση. Στις υπερπεριφερειακές περιοχές θα βρούμε για παράδειγμα την γαλλική Γουιάννα που είναι η μόνη χερσαία περιοχή με σύνορα στη Βραζιλία. Θα βρούμε και το νησί της Ραϊνιόν στον Ινδικό ωκεανό. Θα βρούμε τις νήσους Γουαδελούπη και Μαρτινίκα στις, Καρα... στις Αντίλες. Έχουμε ένα ευρύτατο γεωγραφικό πλαίσιο με τεράστιο δυναμικό Εξάλλου, θα πρέπει εδώ να υπενθυμίσουμε ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι η μεγαλύτερη, έχει τη μεγαλύτερη οικονομική αποκλειστική ζώνη, αυτό οφείλεται στη θάλασσα, στην ωκεάνια περιοχή που έχουν αυτές οι υπερπεριφερειακές περιοχές. Και αν σκεφτούμε τις ισπανικές και πορτογαλικές κτίσεις, στη Μαδέιρα, τα Κανάρια νησιά, τις Αζόρες. Έχουμε μία, την, ε, ε, ε, τα, τα νησιά της, των, της, των Καναρίων που επεκτείνονται πέρα από την Αφρική στον ωκεανό. Αυτό απαιτεί και την διεθνική συνεργασία όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι περιφερειακές περιοχές μπορούν να κερδίσουν πάρα πολλά πράγματα από αυτή την περιφερειακή, διαπεριφερειακή συνεργασία. Και αυτή είναι μια διάσταση που είναι προφανής σε σχέση με την έκθεση που συζητάμε για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Και πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρέπει να μπορέσουμε να υποφεληθούμε από αυτή τη γεωστρατηγική θέση σε σχέση με αυτές τις περιφέρειες. Εδώ υπάρχει μεγαλύτερο δυναμικό ισόρροπων σχέσεων σε σχέση με αυτές τις περιοχές, όπως για παράδειγμα με την ε, περιοχή των ε, Μακαρίων Ίσων, δηλαδή των Κανάριων ε, νησιών ε, και εδώ πρέπει να θέσουμε το κέντρο βάρους στη συζήτηση και να δούμε τους περιορισμούς που είναι παράλογοι καμιά φορά σε σχέση με τη διαπεριφερειακή συνεργασία. Υπάρχει ένα όριο Δηλαδή η απόσταση, μέγιστη απόσταση 150 χιλιόμετρων λέει σε σχέση με την ε, ε, απόσταση, συνοριακή απόσταση. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να κατανοήσω πώς μπορεί να καθορίζεται έτσι το όριο των 150 χιλιόμετρων. Γιατί να μην είναι διαφορετική αυτή η απόσταση. Είναι παράλογο και μ, χαζό να υπάρχει ένα τέτοιο όριο. Απλά καταργεί τις δυνατότητες μιας υπερπεριφερειακής περιοχής να προβαίνει σε διαπεριφερειακή συνεργασία μια και υπάρχει αυτό το όριο. Σήμερα το πρωί σε σχέση με τον Επίτροπο και την παρουσία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα εξεταστεί αυτό, θα εξεταστούν αυτά τα θέματα. Όχι όμως σε σχέση με κάποια κατάργηση, γιατί τίποτα άλλο δεν θα μπορούσαμε να εξετάσουμε, αλλά θα θέλαμε να εξεταστεί και να ληφθεί υπόψη μήπως αυτός ο περιορισμός που δεν έχει κανένα νόημο αν θα μπορούσε να αρθεί, να καταργηθεί και να ανοίξει το δυναμικό που μπορεί να εκμεταλλευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη διαπεριφερειακή συνεργασία. Και θα μπορέσει στο τέλος τέλος ε, να δώσει τη δυνατότητα οι υπερπεριφερειακές περιοχές να ενδυναμώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε θα ήθελα, ο κύριος Ογώ μάλλον, στις υπερπεριφερειακές ζώνες και τα προβλήματά τους. Θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την τύχη χάρη στις υπερπεριφερειακές περιφέρειες να είναι παρούσα σε όλα τα μέρη του κόσμου και συχνάκης να γειτονεύει με μεγάλες αναδυόμενες χώρες. Παίρνουμε πολύ λιγότερο χρόνο, τρεις φορές λιγότερο χρόνο να πάμε τη Ρενιού στην Κίνα από ότι από τη Ρενιού στις Βρυξέλλες. Άρα υπάρχει σημαντική γυτνίαση εκεί που δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη στην ε, πολιτική ε, γειτονία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρησιμοποιεί αυτή τη δυνατότητα, αυτές τις δυνατότητες. Εγώ θα ήθελα, θα ευχόμουν να εκμεταλλευτούμε το ότι οι υπερπεριφερειακές ζώνες είναι τα ενεργά σύνορα, τα δραστήρια σύνορα της ε, Ευρώπης σε όλο τον κόσμο, στο σύνολο του κόσμου. Αν αυτή η πολιτική αρχή εφαρμοστεί, θα ήταν καλό να εφαρμόσουμε την ελόγω πολιτική. Με τα μέσα της πολιτικής ευρείας γειτονίας ε, ή με κάτι άλλο Υπάρχει όμως κάτι που μπορούμε να κερδίσουμε από την Ευρώπη και δεν το χρησιμοποιούμε. Και όχι μόνο από την Ευρώπη και οι άλλες χώρες μπορούν να ωφεληθούν από μια συνεργασία χάνουμε όταν δεν βασιζόμαστε στις περιφερειακές περιοχές. Υπάρχει ένα κενό που καλό θα ήταν να καλυφθεί. Και εφόσον το συζητούμε την ευκαιρία τη εκθέσεως στο ζήτημα, πιστεύω ότι σίγουρα θα πρέπει να φτάσουμε σε μια θετική απόφαση. Δηλαδή ότι αυτές οι υπερπεριφερειακές περιοχές να θεωρηθούν πράγματα σαν ενεργά σύνορα της Ευρώπης στον κόσμο. Euh, euh, θα ήθελα να ρωτήσω τους αγορητές να θέσω κάποια ερωτήματα με θέματα που άπτονται περισσότερο της γυπνιάσεω. Όταν μιλάμε για την εξευρωπαϊκή διεθνή διάσταση περιφερειακής πολιτικής, να δούμε πώς συμμετέχουν και μπλέκονται οι περιφέρειες αυτού του είδους της πολιτικές και τη διάσταση. Και γνωρίζω μάλιστα ότι κάποιες περιοχές όπως η Καταλωνία κάνουν πολλά όσον αφορά την αποκεντρωμένη συνεργασία και ότι αν θέλουμε να προωθήσουμε το μοντέλο της περιφερειακής ανάπτυξης είναι πράγματι αναγκαίο κατά την άποψή μου να το κάνουμε αυτό χρησιμοποιώντας τις περιφέρειες. Έτσι δε περαιτέρω, όταν μέσω της σου όλο και περισσότερο μιλούμε για μακροπεριφέρειες, άλλο επικάλυψη μεταξύ των διαφόρων περιφερειακών πολιτικών που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών ε, των ευρωπαϊκών περιφερειών και των περιφερειών γειτνιάσεως. Πώς διαρθώνονται όλα αυτά. Πώς μπορούν να είναι περισσότερο παρούσες οι ε, περιφέρειες στις πολιτικές που αναφέρονται. Δεν έχουμε άλλους ομιλητές στους ε, καταλόγους. Μπορούμε να επεκτείνουμε τα θέματα αυτά και στην πολιτική γυτνιάσεως. Λοιπόν, όποια σχόλια έχετε θα σας είμαι θα ευγνώμονες να τα ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Καταρχάς, όσον αφορά... Α, αυτό που έδειξα είναι ένα γενικό φυλάδιο. Δεν είναι μια έκθεση που αναφέρεται στα πεπραγμένα των περασμένων ετών. Μπορούμε να σας δώσουμε επίσης και άλλες πληροφορίες που δίνουμε προφανώς στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, για να δείξουμε πώς εφαρμόζουμε όλα αυτά τα μέτρα. Μπορούμε να σας αποστείλουμε στη γραμματεία τα σχετικά έγγραφα και τις πληροφορίες. Τώρα, για να σας διαβεβαιώσω πόσο καλά τα πήγαμε πέρσι. Δίκιο έχετε με αυτά που είπατε ότι είναι πολύ δύσκολο, δύσκολα πράγματα. Είναι απρόβλεπτος ο φόρτος εργασίας και ακόμα και όταν θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ καλό το προϊόν μας, όπως είπατε κύριε Βανίστερ Ρόι, στην κοινή έκθεση. Θέλαμε να ασχοληθούμε με την Κίνα, με, με τη συνεργασία του ΟΣΑ, στην περιφερειακή καινοτομία. Και στο τέλο οι Κινέζοι είπαν όχι, δεν θα πάρουμε. Δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα. παρόλα αυτά, στο τέλο του έτου είχαμε 85%, ε, ανάληψη υποχρεώσεων από τα χρήματα που έχουν διάθεσή μα. Είναι μεγάλη πρόκληση για μα, σωστά το λέτε, δεν έχουμε και άλλου πόρου. Είναι δύσκολο να χειριστούμε αυτό το προϊόν και μέσω της δράσεως αυτής να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα στην πραγματικότητα. Αναφέρατε και σε ευχαριστώ για αυτό ότι η επόμενη συνάντηση υψηλού επίπεδου για την περιφερειακή πολιτική Ευρωπαϊκής Ενώσεως Κίνας ε, θα είναι στις 30 Οκτωβρίου στα Open Days και στις 13 Οκτωβρίου. Λοιπόν, τονίσαμε ότι είναι πολύ τιμή η υποστήριξη που μας παρέχεται. Προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού να συνδυώσουμε τους διάφορους πόρους. Στην περίπτωση της Ρωσίας, η βασική που χρησιμοποιούμε δεν είναι από τα πιλωτικά προγράμματα, αλλά περισσότερα από το μέσο υποστήριξης που υπάρχει στα πλαίσια των εξωτερικών σχέσεων. Στην περίπτωση της Βραζιλίας, η Βραζιλία μάλλον, είναι ο βασικός ετών για την χρήση του μέσου για την υποστήριξη διαφόρων συζητήσεων και διαλόγων. Σωστά αναφέρεται το ρόλο των υπερπεριφερειακών περιοχών που είναι στην πρώτη γραμμή. Στόχος μας είναι να συμμετάσχουν όσο δυνατόν περισσότερες περιφέρειες. Ξεπερνώντας και τα όρια των υπερπεριφερειακών περιφερειών. Ανέφερα φέτος τον Οκτώβριο τι θα γίνει. Θα πάνε, κάποιοι Μολδαβοί θα πάνε στη Λετωνία, Γεωργιανοί θα πάνε στην Ισπανία κλπ. κλπ. Θα γίνονται επισκέψεις. Τονίσαμε ότι είχαν προνομιούχες σχέσεις με τις υπερπεριφερειακές ζώνες. Κυρίως με τη Γαλλική Γουιάννα, όπω είπατε κύριε Ντεξέρα. Δεν, δεν, δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για την ομορφιά τη συνοριακή συνεργασία στην Λατινική Αμερική και στο επίκεντρο είναι η Βραζιλία που γειτονεύει με όλε τι χώρε εκτός από δύο στην Λατινική Αμερική. Άρα χρειαζόταν και κοινό προγραμματισμό με τη Γαλλία λόγω τη Γαλλική Γουιάννα και μαζί με το Σουρινάμ. 100% σχεδόν ανάληψη υποχρεώσεων είχαμε σε αυτά τα προγράμματα. Δώσαμε νέα όθηση λοιπόν. Και φαινόμενο μόχλευσης και σε εθνικό επίπεδο. Είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με δυτικοαφρικανικές χώρες. Μακαρονισία, Κανάρι, Νήσι, είμαστε κοντά στη Σενεγάλη, υπάρχουν και πολιτικά συμφέροντα εκεί. Δεν μπορέσαμε να τους δώσουμε κίνητρα όμως να είναι πιο ενεργοί. Οι συνάδελφοι που είναι υπεύθυνοι για τις υπεραπομακρυσμένες περιοχές ίσως μπορούν να βοηθήσουν να δουν πώς να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δράσεις, το διάλογο για να προωθήσουμε τον προνομιούχο ρόλο των υπερπεριφερειακών ζωνών. για το ερώτημα του κύριου Αλφόντσι. Δεν έχουμε δυνατότητα να να συντονίσουμε τις προσπάθειες που έχουν δρομολογηθεί και τις άμεσες επαφές μεταξύ περιφερειών ευρωπαϊκών και διαφόρων περιφερειακών, περιφερειών εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Μπορούμε όμως να εκμεταλλευτούμε μέσω οργανώσεων μελετών των εκπροσώπων τους, αλλά και αναφέροντας και τις δραστηριότητε που έχουν αναλυφθεί. Στις Open Days θα έχουμε επισκέψη του Υπουργού Διεθνούς Συνεργασίας της Βραζιλίας και θα έχουμε μία δράση των τεσσάρων κινητήρων που έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συντονιστούμε στις τέσσερις κινητήρες που χρησιμοποιούν ε, για τις προσπάθειες αυτές στη Λατινική Αμερική. Θέλουμε να συμμετάσχουν διάφοροι εμπλεκόμενοι, ευρωπαϊκές ενώσεις των παραμεθεριών περιφών, διάφοροι φορείς. Όλοι μαζί να έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο σε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Δεν έχουμε όλους τους πόρους που απαιτούνται να συντονίσουμε τα πάντα. Και τις, να συντονίσουμε και όλες τις δράσεις που γίνονται πολύ σωστά από τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Αν δεν υπάρχουν σχόλια όσον, ε, όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος Γκουλέ, μπορούμε να προχωρήσουμε στην παρουσίαση. Ο κύριος Όλμπρεχτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Έχω την εντύπωση, εντάξει, μπορώ να κάνω λάθος, ε, αλλά αυτό αποτελεί πολύ καλό παράδειγμα της ε, συντονισμού από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί έχουμε την Επιτροπή ανάπτυξη, την Επιτροπή Περιφερειακής ανάπτυξη. ε, και από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε πολλά κοινά ζητήματα στα οποία συνεργαζόμαστε μεταξύ των δύο, οι δύο αυτές επιτροπές. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούν αυτές οι δύο επιτροπές. Κοιτάζω τα έγγραφα που προετοίμασε η Επιτροπή Ανάπτυξης και δεν υπάρχουν ε, σχεδόν καθόλου στοιχεία περιφερειακής πολιτικής που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την αναπτυξιακή πολιτική. Ένα άλλο παράδειγμα. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για το διεθνές σκηνικό είναι το ζήτημα των αστικών κέντρων. Ε, μέσα στην ομάδα μου με τους αδέλφους μου εντοπίσαμε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον σε παγκόσμια κλίμακα για την ευρωπαϊκή εμπειρία στην ε, αναζωογόνηση των αστικών κέντρων και πιο συγκεκριμένα του χρόνου θα διεξαχθεί το Διεθνές Φόρουμ Αστικών Κέντρων στην Άπολη. Και ξέρω ότι αυτό το Διεθνές Φόρουμ βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μας ζήτησαν να συνεργαστούμε μαζί τους για να προετοιμάσουμε ένα μέρος ε, του συνεδρίου, δηλαδή να ε, μοιραστούμε την εμπειρία μας σε ό,τι αφορά την ε, αστική πολιτική, τμήμα δηλαδή της περιφερειακής πολιτικής. Ξέρουμε ότι υπάρχει δυσκολία σε αυτόν τον ορισμό μεταξύ περιφερειών και πόλεων, αλλά και πάλι θα είναι ένα χρήσιμο, μια χρήσιμη εμπειρία ε, τονίζοντα ιδιαίτερα την ε, σημασία της περιφερειακής πολιτικής. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή θέλει να απαντήσει. Όχι. Θα πρέπει να επανέλθουμε στο ζήτημα το οποίο θίξατε, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο εμά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ διαφόρων επιτροπών. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την συνεργασία των ε, ε, επιτροπών. Όχι μόνο με την Επιτροπή Ανάπτυξης, αλλά και με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Το, τα ζητήματα γυτνίασης είναι θεμελιώδης σημασία για όλες αυτές τις επιτροπές του Κοινοβουλίου, για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις προκειμένου να ανοίξουν έγγραφα, παραρτήματα, δεν ξέρω πώς τα λένε, κανονισμοί που αφορούν τις ε, αρμοδιότητες των ε, Επιτροπών του Κοινοβουλίου. Πρέπει όμως να δούμε τι θα κάνουμε χωρίς ε, να αλλάξουμε τον ιστορικό κανονισμό ε, του Κοινοβουλίου. Χωρίς να αλλάξουμε λοιπόν κάτι, πώς μπορούμε να γίνουμε πιο ευέλικτοι. Λάμπερτ. Το πυροτικό σχέδιο, από ό,τι κατάλαβα, δίνει μια περαιτέρω δυνατότητα ανταλλαγής, συνεργασίας με τους Ευρωπαίους εταίρους ε, για την ε, πολιτική συνοχή μας. Και αυτό αφορά συγκεκριμένε χώρε όπω η Βραζιλία, οι χώρε τη Αφρική και το καθεξή. Όμω αυτό αφορά και μια πολιτική. Και η πολιτική δεν είναι πιλωτικό σχέδιο. Το πιλωτικό σχέδιο είναι κάτι πιο περιορισμένο. Αν κατάλαβα καλά την Επιτροπή. Όμω, η ίδια πολιτική είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε. Τώρα έχουμε την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γετνίασης. Τώρα εξετάζεται από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και από όσο ε, βλέπω η πολιτική γετνίαση αλλάζει. Μεταμορφώνεται και ε, λαμβάνει το χαρακτήρα μη κυβερνητικής ε, συνδρομής στην διαδικασία εκδημοκρατισμού και ούτω καθεξής. Ίσως λοιπόν είναι φρόνιμο ε, να κάνουμε αυτό τον διάλογο τώρα. Δηλαδή ποια εργαλεία είναι πραγματικά αποτελεσματικά στην ε, περιφερειακή πολιτική και στην διασυνοριακή συνεργασία. Και ποιοι είναι οι περιορισμοί μας. Αυτά τα 150 χιλιόμετρα και ούτω καθεξής. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Αλλά ας πούμε για του χρόνου. Όταν θα ξανάρθετε και θα κάνετε μια νέα παρουσίαση, να δούμε αν θα έχουμε νέα στοιχεία από την ευρωπαϊκή ε, πολιτική σας. Γιατί εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Ε, ε, χάνουμε το στόχο μας αν βασιζόμαστε μόνο στις πρωτεύουσες για να καθορίσουν τις πολιτικές. Έχουμε τόσες δυνατότητες να αξιοποιήσουμε τα, τα πολύ αποδοτικά αυτά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα. Εργαλεία τα οποία λειτουργούν σε διασυνοριακό επίπεδο. Και στηρίζω τον συνάδελφο Γιάννη Όλμπινγκ. Έχουμε εδώ πολιτικές, πολιτικές ανάπτυξης, πολιτικές ε, εξωτερικών υποθέσεων. Αλλά εγώ, α πούμε, ζήτησα τι, στην ε, ΑΦΕΤ, τι κάνετε με τα σύνορα. Έχουμε όλο αυτό το σχεδιασμό για την πολιτική γυτνίαση, αλλά στο τέλος τι απομένει από την ε, συνεργασία. Συμφωνώ λοιπόν απολύτω με τον Γιάννη σε αυτό που είπε για τις πόλεις, για τα αστικά κέντρα. Ίσως αυτή θα ήταν η απάντηση, ε, να συμπεριλάβουμε δηλαδή για τις πόλεις το 2012. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον Πίτε Μπέρκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πολύ σύντομα θα παρουσιάσω μία ε, μελέτη την οποία ε, εκπονήσαμε εμείς ε, για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχή σε παγκόσμιο επίπεδο ή σε σφαιρικό επίπεδο. Την ανέλαβε η σε σφυρικο επιπεδο την Διεύθυνση ε, Περιφερειών και επικεφαλής ήταν ο Τζον Ε, Στόχος ήταν να ε, συγκρίνει την πολιτική συνοχή με άλλες ε, πολιτικές ε, που χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα κοινής διαχείρισης, επιμερισμένης διαχείρισης. Συλλέξαμε στοιχεία από χώρες ως αλλά και διεθνείς δημοσιονομικούς οργανισμούς. Και τέλος ε, θέλαμε να εντοπίσουμε συγκεκριμένα και να αντιλήσουμε μαθήματα για την ε, πολιτική αυτή. Βασίστηκε σε ε, περιπτωσιακές μελέτες και studies που αφορούν χώρες του ΩΣΑ αλλά και ευρωπαϊκές χώρες αλλά και από διεθνείς οργανισμούς όπως τον EBRD και την Παγκοσμία Τράπεζα. Κίνητρο για αυτή τη μελέτη ήταν το ότι στη συζήτηση για την πολιτική συνοχή πολύ συχνά Ακούσαμε τι θα έκαναν άλλες χώρες ή άλλοι οργανισμοί. Δεν, υπήρξαν, ε, δεν υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία συγκριτικά. Βάσει όμως του έργου που κάνουμε με τον ΩΣΑ, αλλά και τη συνεργασία μας με, το, με την Παγκόσμια Τράπεζα, καταλήξαμε σε αυτή τη μελέτη. Είναι πολύ πλούσια αυτή η μελέτη, δεν έχω πολύ χρόνο, έτσι σας καλώ να την εξετάσετε σε βάθος. Θα ήθελα όμως ε, να αναφερθώ σε ορισμένα από τα βασικά συμπεράσματα ε, στα οποία καταλήξαμε με βάση αυτή τη μελέτη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Η μελέτη αυτή λοιπόν εξέτασε τι συμβαίνει σε άλλες χώρες με ομοσπονδιακά συστήματα, τι γίνεται με τις ε, περιφέρειές τους και, και πάντα σε σχέση και με οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα. Η πρώτη σύσταση που προκύπτει από αυτή τη μελέτη είναι ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, σχέση μεταξύ του κέντρου, στην προηγούμενη περίπτωση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Ίσως να υπάρχει και ένα συμβατικό πλαίσιο. Αυτό το καλούμε εμείς ε, εταιρική σχέση, partnership contract, σύμβαση εταιρική σχέσης. Όμως αυτό απαιτεί περαιτέρω πόρους. Όταν αλλάζουμε τη δομή και την σύνδεση μεταξύ των δύο μερών, αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τους απαραίτητους πόρους για να το κάνει αυτό, αλλά το ίδιο ισχύει και για τις περιφέρειες και τα κρατημέλη. Μία σύσταση είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση των δημοσιονομικών εργαλείων βάσει εμπειριών από ε, το εξωτερικό, αλλά πάντα συνιστάται και προσοχή. Για να δουν δηλαδή τα κρατη και επιτροπή το πού χρησιμοποιούν άλλα εργαλεία, πού χρησιμοποιούν δανεισμό και μόχλευση για να ε, λαμβάνουν υπόψη και το, τις περιπτώσεις στις οποίες αυτά είναι, τα εργαλεία είναι πιο αποδοτικά. Ε, εστιάζει επίσης η μελέτη στους όρους και τις προϋποθέσεις, αλλά και την πολυπλοκότητα αυτών. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι δύσκολο να συνάξουμε συμπεράσματα βάσει των δεδομένων για το τι είναι αποδοτικό και τι όχι όταν αλλάζει από το ένα πλαίσιο και πας στο άλλο. Ε, δίνεται εντύπωση ότι, αυτό που κάνουμε εμείς ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, ήδη μας δίνει ένα τέτοιο, μια εικόνα αυτών των όρων υπερποθέσεων. βεβαίως αυτό ισχύει και σε άλλες πολιτικές και ενώ η πολιτική συνοχή δεν έχει συγκεκριμένες περιποθέσεις προς το παρόν. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτό το επίπεδο. Γενικά η μελέτη στηρίζει στηρίζει την ε, περαιτέρω χρήση αυτής της αιρεσιμότητας, αλλά εστιάζει σε διάφορες ε, μορφές ε, εκ των προτέρων ερεσιμότητα ε, που συνδέεται με την διαχείριση, διακυβέρνηση και ούτω καθεξής. Κυρίως όμως ε, εστιάζουμε τι συμβαίνει σε μακροφορολογικό επίπεδο. Εστιάζει, ε, τονίζει μάλλον τις θετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά ε, εφιστάκεται την προσοχή ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ορισμένες μορφές κοινωνική πολιτική, για παράδειγμα κοινωνικού στόχους και υπάρχει και το θέμα του ποιο είναι υπεύθυνο. Και αυτή η πτυχή για την εφαρμογή αυτών των ερησιμοτήτων. Δηλαδή, ορισμένε φορέ οι κυρώσει επιβάλλονται όσου δεν, δεν ήταν υπεύθυνοι για την λήψη τη απόφαση. Η μελέτη ε, συμφωνεί και στηρίζει την ύπαρξη ερεσιμοτήτων που ε, συνδέονται άμεσα με την ενίσχυση της αποδοτικότητας ε, των πολιτικών βάσει και ε, παραδειγμάτων που έχουμε δει από αλλού για την ερεσιμότητα βάση επιδόσεων. Πάντα στο πλαίσιο της βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ κέντρου και περιφερειών. Ε, θα πρέπει να εστιάσουμε και την θεσμική στήριξη για την ε, διακυβέρνηση του δημοσίου τομέα. Η μελέτη λοιπόν αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη συζήτηση ε, και εδώ στο ιστορικό του Κοινοβουλίου αλλά και μεταξύ ενδιαφερομένων μερών. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο σαφές συμπέρασμα ακόμα. Μετά προχωράμε στα κίνητρα και τις χειρώσεις πάλι βασίζεται σε, στην εμπειρία σε άλλα μέρη του κόσμου για τα κίνητρα και τις ε, κυρώσεις και υπογραμμίζει ότι υπάρχουν λιγότερες κυρώσεις στην πολιτική συνοχή σε, σχέση με τα IFIs και το γεγονός ότι έχουμε αυτά τα, τα εργαλεία ευρείας ε, βάσεως ε, καθιστά πιο δύσκολη την χρήση τους στο πλαίσιο ενός συστήματος κυρώσεων. Γιατί εξάντε πρόκειται για ένα σύστημα κατανομής ε, πόρων. Τώρα, βάσει της ε, εμπειρίας που λαμβάνουμε από εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτον οι κυρίες πρέπει να είναι αναλογικές. Δεύτερον, υπάρχει το θέμα της, ε, ε, του ρόλου του ιδιοκτήτη ή του δικαιούχου ε, στην κατάσταση που μπορεί να επιφέρει επιβολή κύρωσης. Και δεύτερον, το ζήτημα μιας βαθμιαίας μάλλον προσέγγισης. Η μελέτη στηρίζει την ευαρξή κινήτρων και βάση επιδόσεων ενδεχομένως, αλλά ε, από μεθολογικής άποψης μπορεί να, υπάρχουν, να αποτελέσει αυτό πρόκληση. Τώρα περνάμε στην αξιολόγηση. Καταλήγουμε σε δύο συμπεράσματα. Πρώτον, ότι υπάρχει ένα πεδίο εφαρμογή, αν θέλετε, ένα ε, σκοπό για την ύπαρξη αυτή τη αξιολόγηση. Αλλά ε, πρόκειται για μια πολιτική η οποία έχει αξιολογηθεί πολλάκι. Επομένω, το θέμα δεν είναι να καταλήξουμε σε ένα νέο σύστημα, αλλά να βελτιώσουμε το υπάρχον σύστημα μέσω των αξιολογήσεων. Υπάρχουν και ορισμένε ε, μορφέ ε, και μεθοδολογίε, για παράδειγμα στην Παγκόσμια Τράπεζα, οι οποίε ενδεχομένω να μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ε, για τη δική μα πολιτική. Τέλο, η μελέτη εξετάζει και πρότυπα αξιοπιστία. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πρότυπα το πρότυπο το οποίο ε, αξιοποιούμε εμείς στην πολιτική συνοχής αποτελεί, ανήκει στην μια, ειδική κατηγορία, θέλετε, στη δική του κατηγορία, είναι sui generis, βασίζεται στην κατανομή των, ε, των αποδοχών περισσότερο όμως ε, δεν κάνουμε συστάσεις σε αυτό το τομέα. Βεβαίως υπάρχει ε, ανάγκη απλούστευσης, ε, διευκρινήσεων, κατάρτισης, να εστιάζουμε περισσότερο σε μια προσέγγιση ανάλογα με τους κινδύνους, αναλογικότητα πάντα στους ελέγχους και στις προϋποθέσεις ελέγχων. Το γενικότερο μήνυμα όμως ε, το οποίο αντιλήσαμε από εδώ είναι ότι βρίσκουμε στοιχεία που στηρίζουν τις ιδέες που έχουμε υποβάλει και παρουσιάσει και που συζητούνται για το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής. Ταυτόχρονα όμως η μελέτη υπογράμμισε το γεγονός ότι δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τα ίδια συστήματα από τον ένα τομέα στον άλλον. Μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε τέτοιε περιπτώσει. Και τέλος, αν και δεν πρόκειται για άμεσο συμπέρασμα της μελέτης, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η πολιτική συνοχή ήδη λειτουργεί και έχει αποτελέσματα. Βεβαίως πολλά μπορούν να βελτιωθούν, αλλά έχουμε μια καλή βάση. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις όσον αφορά την παρουσίαση αυτή την χρονική στιγμή, την χρονική συγκυρία δεν υπάρχουν. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πω ότι όλες αυτές οι μελέτες και οι πληροφορίες που παρουσιάσατε είναι διαθέσιμες, αλλά μπορείτε να αποστείλετε κάτι και ηλεκτρονικά στη γραμματεία μας και έτσι μπορούν να διανεμηθούν ατομικά και αυτά τα στοιχεία θα ήταν πραγματικά θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας διανύμετε, να μας αποστείλετε τέτοιες πληροφορίες. Μπορούμε να κλείσουμε νομίζω εδώ αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Και έτσι από πλευράς ε, του εκπροσώπου Μίχαηλ Τόρερ που βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω σε σχέση με τους σκιώδεις. Ε, ο Πέτα Ζήμερ δεν παρίσταται. Όμως ο Μιχαήλ είναι εδώ παρόν. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον Μιχαήλ, με την παρουσίαση λοιπόν του Μιχαήλ Τόερα για την, α, απόψεις για την ευρωπαϊκή πολιτική και την, είναι γνωμοδότηση της Οικονομικής Νομισματικής Επιτροπής ΕΙΚΟΝ. Μιχαήλ Τόερα, έχετε τον λόγο λοιπόν τώρα παρακαλώ. Μάλιστα, yeah. σας ευχαριστώ αξιότιμε πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ασχολούμαστε σήμερα με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δραστηριοτήτων υπό το πρίσμα της πολιτικής συνοχής. Πρώτα απ' όλα καταρχήν συμβαίνει το εξή. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο εισάγεται, εισήχθη σαν συνέπεια και συνέχεια των μέτρων για την υπέρβαση και αποφυγή μελλοντικών ευρωκρίσεων και της κρίσης της ε, κρατικής υπερχρέωσης από τα κράτη-μέλη. Είναι μια περαιτέρω εξέλιξη, η μεταξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να συναρθούν τα συμπεράσματα και διδάγματα, οι διδαχές από την κρίση και κρίση υπερχρέωσης στην Ευρώπη. Οι Υπουργοί Οικονομικών ε, ε, το Σεπτέμβριο 2010 αποφάσισαν να ξεκινήσει αυτό το Ευρωπαϊκό εξάμεινο. Η διαδικασία προβλέπει ότι την μακροπρόθεσμη, το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του στα κράτη-μέλη έγκαιρα θα τον γνωστοποιούν στις Βρυξέλλες. Μετά από μια τέτοια γνωμοδότηση θα εγκρίνονται οι προϋπολογισμοί των κρατών μελών. Είναι μια προληπτική εποπτεία των προϋπολογισμών τους δημοσιονομικά μέσα στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ώστε οι αρχές να μπορούν, οι αρχές για αυτή την πολιτική να εφαρμόζονται. Έχουμε λοιπόν εδώ και τα θέματα των μακροοικονομικών ανισορροπιών και για τον σχεδιασμό που πρέπει έγκαιρα να αναγνωρίζονται και να αποφεύγονται. Και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική Πειθαρχία και Δημοσιονομική Πειθαρχία, θα πρέπει να εντάσσεται και να προαγάγει την πολιτική για την Ευρώπη 2020. Πρόκειται για δική μας γνωμοδότηση που διαβιβάζουμε στην αρμόδια επί της ουσίας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Πρόκειται για ένα αποτελεσματικό μέσο για την υλοποίηση της στρατηγικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2020. Και κατά τούτο η πολιτική συνοχή διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο. <clears throat> Μια ισχυρή και παγιωμένη πολιτικής συνοχής μπορεί και μακροπρόθεσμα στα αναπτυξιακά προγράμματα μέσω της αποκεντρωμένης ε, διοίκησης και με θέσπιση προτεραιοτήτων από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει στην αηφορία της ανάπτυξης και να είναι μια σημαντική οικονομική προώθηση της πολιτικής. Και αν γίνει σωστή, σωστά αυτή η εφαρμογή μπορεί να είναι μια σωστή ε, συνεισφορά για την μακροοικονομική ισορροπία. Κατά τούτο πιστεύω εγώ ω εισηγητής ο συντάκτη νομοδότησης ότι αξίζει τον κόπο να προβληματιστούμε σε αυτό το πλαίσιο και να δούμε τι μπορεί να γίνει σε σχέση και με προτινόμενες κυρώσει και τι μπορούμε να κάνουμε όταν κράτη δεν τηρούν την πειθαρχία όσον αφορά τα θέματα της ε, υπερχρέωσης αν έχει κάποιο νόημα να περικόπτουμε κονδύλια των διαθετικών ταμείων ή των περιφερειακών ταμείων ή αν θα πρέπει να έχουμε αντίθετα κίνητρα ένα σύστημα ας το πω έτσι σταθεροποιητικών μέτρων που στην κρίση που διανύουμε Τώρα για παράδειγμα η Ελλάδα αν μπορεί να συνεισφέρουν αυτά τα μέτρα ώστε να επιστρέψουμε σε μια οδό, μια πορεία ανάπτυξης ε, και απασχόλησης. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο λοιπόν είναι μια πρόοδος όσον αφορά τον συντονισμό στο οικονομικό επίπεδο και σίγουρα εδώ έχουμε ένα σε, πολλές, ε, σε πολλά βήματα κλιμακούμενο πρότυπο η περιφερειακή πολιτική έχει ήδη μια παγιωμένη μέθοδο, μεθοδολογία όσον αφορά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και προσφέρει ένα σωστά ισορροπημένο ε, φορολογικό σύστημα επιτόπου ή φορολογική πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις μέσα στο πλαίσιο των διαθροτικών πολιτικών ή και μάλιστα ότι δεν είναι αναγκαίες τέτοιες διαθροτικές ε, προσαρμογές και αλλαγές, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε σε τέτοιο πλαίσιο, μια και σήμερα έχουμε να συζητήσουμε για την ε, πολιτική συνοχή και να δούμε και το θέμα της απορροφητικότητας, του ποσοστού απορροφητικότητας που και εδώ διαδραματίζει και αυτό ένα ρόλο. Εν πάση περιπτώσει, οπωσδήποτε, τα διαθωτικά κονδύλια, τα διαθωτικά ταμεία διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Είναι μια σημαντική συνεισφορά ώστε η έρευνα, η ανάπτυξη, η καινοτομία στο εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο να μπορέσουν να προαχθούν και να δράσουν σωστά. Κέντρα βάρου, εν πάση περιπτώσει, είναι εμείς διαπιστώνουμε ότι οι εθνικοί στόχοι εν μέρη δεν είναι υπερβολικά φιλόδοξοι όσον αφορά το πλαίσιο της στρατηγικής 2020 φαίνεται εδώ να υπάρχει μια αιμονή σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα σε σχέση με μια μακροπρόθεσμη, αν θέλετε, ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα αηφορίας, κοινωνικής συνοχής ε, και περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας. Απέχουμε ακόμα σε σχέση με τους στόχους ε, του 2020, της στρατηγικής για το 2020, απέχουμε πολύ πόρο απέχουμε από το να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι. Εδώ λοιπόν η διαθροτική πολιτική θα συνεισφέρει. Η κατεύθυνση στην διαθροτική πολιτική πρέπει να έχει τέτοιο, τέτοια μορφή ώστε το περιφερειακό δυναμικό να τονωθεί και να λαμβάνεται υπόψη ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Κατά τούτο, η διαθροτική πολιτική μπορεί να συνεισφέρει από πλευρά τη ώστε η Ευρώπη επιτόπου στι περιφέρειε, στα αστικά κέντρα τη πόλη, αλλά και στι κοινότητε και του Δήμου να διαδραματίσει ένα ρόλο για την υλοποίηση των στόχων και τη στρατηγική σε όλα τα επίπεδα, όπω απαιτείται. Έτοιμα είναι τα κράτη-μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια, οι κοινωνικοί εταίροι, οι περιφερειακέ και τοπικέ αρχέ, αλλά και οι επιχειρήσει και η κοινωνία των πολιτών να εμπλακούν στενότερα εκ του σύνεγγυς στη διαμόρφωση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης και αναθεώρησης, ώστε να υπάρξει και μια σε τακτά διαστήματα ε, δυνατότητα διαβούλευσης και συντονισμού. Αυτά είναι τα ουσιοδέστερα στοιχεία εν συντομία του σχεδίου γνωμοδότησής μου. Χαίρομαι για τη συζήτηση αυτών των ε, προτάσεων και θα περιμένω να ακούσω τα σχόλιά σας και τις τροπολογίες σας ώστε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία ώστε οι θέσεις που από κοινού εκπροσωπούμε στην Επιτροπή να τονιστούν ιδιαίτερα και να καταστούν σαφέστερες, διότι η πολιτική για τη συνοχή έχει μια υποτιμημένη σπουδαιότητα και σημασία για την μακροοικονομική σταθεροποίηση και την επιστροφή στην οδό της απασχόλησης και ανάπτυξης, ιδιαίτερα για χώρες ε, που έχουν πληγεί και έχουν, ε, φέρουν βαρέως την κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μικαέλ. Κυρία Κράτσο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την παρουσίαση που μας έκανε, καταρχάς ως προς τη σημασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πράγματι, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι μια νέα παράμετρο συμπλήρωσης του πακέτου οικονομικής διακυβέρνησης και συμβάλλει ως προς την ενίσχυση του προληπτικού σκέλους ε, των δημοσιονομικών ανισορροπιών ε, και της αστάθειας που έχουμε σήμερα ε, και από την άλλη πλευρά για να εμπεδοθεί καλύτερα η συνεργασία εθνικού και ευρωπαϊκού επίπεδου ως προς τους στόχους και ως προς τις εκτελέσεις των προϋπολογισμών. Τώρα ερχόμαστε εμείς με τη γνωμοδότησή μας να δώσουμε μια διάσταση περιφερειακή. Ε, πιστεύω ότι δύο είναι τα σημαντικά θέματα. Από τη μια μεριά πρέπει στα ευρωπαϊκά εξάμεινα, δηλαδή στους προϋπολογισμούς που καταθέτουν τα Εθνικά Κοινοβούλια να υπάρχουν με σαφήνεια οι στόχοι της συνοχής και θέλω να πω ότι στις συστάσεις που έδωσε προς τα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ δύο εβδομάδων έχει σημασία να το τονίσουμε αυτό, ότι πρέπει να εστιάσουμε ε, περισσότερο σε στόχους και δράσεις που ενισχύουν τη συνοχή. Απ' την άλλη πλευρά είναι πολύ Αυτό σημαίνει ότι τα... οι, τοπικές και οι περιφερειακές αρχές πρέπει να έχουν ένα ε, να ζητήσουμε ένα θεσμοθετημένο διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια για να, μπορούμε, για να ξέρουμε ότι αυτά τα οποία έρχονται ως προτάσεις ε, προϋπολογισμών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη-μέλη έχουν λάβει υπόψη τους τις ανησυχίες και τις θέσεις των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για κάποια κράτη, ε, διότι, τα οποία δεν ε, ε, έχουν αρμοδιότητες μεγάλες στις περιφερειακές αρχές, δεν είναι ίδιο το σύστημα στην Ευρώπη, οπότε έχει σημασία να το τονίσουμε ότι πρέπει να είναι εμπλεγμένα ουσιαστικά στη διαμόρφωση αυτών των προϋπολογισμών. Από την άλλη πλευρά, παίζει ρόλο να συνειδητοποιήσουμε ότι πολλές ανισορροπίες δημοσιονομικές σήμερα οφείλονται σε γκρίζε ζώνες, όπως το χρησιμοποιώ στη χώρα μου, το φέρω και εδώ, γκρίζε ζώνες που είναι από την τοπική αυτοδιοίκηση. Σε εμά, ας πούμε, ε, ε, στην Ελλάδα, μια και αναφέρθηκε και ο συγητής στην Ελλάδα, ε, πολλές, πολλά ε, πολλές πηγές ε, των κακών δημοσιονομικών μας είναι, προέρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι δεν είναι μόνο ο ρόλος των τοπικών περιφερειών ε, για των τοπικών αρχών σημαντικός για, την, για το αναπτυξιακό πρόγραμμα αλλά και για τη δημοσιονομική πειθαρχία που σήμερα είναι ένα μια, μια μεγάλη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα σημειώσει μια απορία, αλλά την έλυσε ο εισηγητή με την παρουσίασή του. Τι εννοεί φιλόδοξου στόχου. Το προσδιορίσατε τώρα, ότι εννοείται ε, στόχους που, στοχεύουν ακριβώς, που αναφέρονται ακριβώς στο Ευρώπη 2020. Ε, αυτό που ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι πρέπει να αναδείξουμε και το ρόλο που πρέπει να παίξει η Επιτροπή Περιφερειών. Είναι ένα όργανο αναβαθμισμένο και από τη συνθήκη της Λισαβόνα και δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία να το εμπλέξουμε ε, και σε αυτή τη διαδικασία και, στον, και στο προληπτικό, στο σκέλος, στο σχεδιασμό και στον απολογισμό που κάνουν ως προς τη συμμετοχή των ε, περιφερειών στα διάφορα κράτη-μέλη. Αυτές είναι τις γενικές γραμμές οι παρατηρήσεις, ε, κυρία Πρόεδρε, και θα δω πόσο μπορώ να τις αποτυπώσω με τις τροπολογίες ε, για την, ε, ε, από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πέτερ Σήμερα παρακαλώ. Τέλεια με την χρονική σας αυτή, το χρονικό σας συντονισμό. Καθίστε και πάρετε τον λόγο παρακαλώ. I'm so sorry if I was in time, but you have been so early. Ε, φτάσατε τόσο νωρί. Συγγνώμη που έφτασα καθυστερημένος. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μίχαλ, για την παρουσίαση αυτή τη γνωμοδότηση. Σε δύο σημεία είχα σκεφτεί και προβληματιστεί αν ίσω όλα αυτά υπό το πρίσμα της δικής μας Κοινοβουλικής Επιτροπής θα έπρεπε να ενταθούν, να ενδυναμωθούν περισσότερο. Το πρώτο αφορά το σημείο 2, το εδάφιο 2. Το θέμα, το ερώτημα, αν μήπως εδώ στις συστάσεις δεν θα έπρεπε να συντάξουμε και να πούμε ότι τα λειτουργικά προγράμματα στις συστάσεις που διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τα λειτουργικά προγράμματα των διαθροτικών ταμείων θα πρέπει να μπορέσουν να λειτουργήσουν να, ε, στοχοθετημένα. Αν τα διαδοτικά ταμεία δηλαδή θα μπορούσαν να είναι ένα μέσο ώστε οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να ε, μπορούσαν να εφαρμοστούν καλύτερα. Ένα δεύτερο σημείο που σε αυτό το σημείο προβληματίστηκα και σκέφτηκα ότι θα έπρεπε ίσως να συζητήσουμε είναι το μήπως θα έπρεπε να είμαστε πιο αυστηροί στη διατύπωση του σημείου 6 στο οποίο ζητείτε τα εθνικά κοινοβούλια, οι κοινωνικοί εταίροι, οι τοπικέ αρχέ κτλ, κτλ, Όλοι αυτοί να εμπλέκονται, να συνεμπλέκονται και να συμμετάσχουν. Αλλά και εδώ είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί. Μια και έχει δικά του ξεχωριστά αιτήματα ω προ αυτό το αίτημα. Ακριβώ για την αρμοδιότητα τη δική μα Κοινοβουλευτική Επιτροπή και την αξιολόγηση άλλων πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την κοινωνική και οικονομική συνοχή. Αν δούμε πώς θα πρέπει τα κράτη να υλοποιούν τις πολιτικές τους συσχετίζεται άμεσα με τα αιτήματά μας. Γι' αυτό θα ήθελα να προβληματιστούμε σε αυτό το σημείο να δούμε, να συμπληρώσουμε ίσως αυτό το σημείο με τα δικά μας αιτήματα, ώστε να συμπεριληφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακριβώς και οι κοινοβουλευτικές του επιτροπές σε αυτό το έργο. Κύριε Τρεμόπουλος, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τόιρερ για το σχέδιο γνωμοδότηση. Οι προτάσει τη επιτροπή μα στην αντίστοιχη αρμόδια Επιτροπή των Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ε, με βρίσκουν σύμφωνο. Ειδικά η παράγραφος 4, ε, όπου γίνεται λόγος για την ανάγκη ενίσχυσης του δυναμικού και των φορέων των περιφερειών, καθώς και στην παράγραφο 6 όπου η συνεργασία των κρατών μελών με τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές κρίνεται ως ανεπαρκής. Έμεσα βέβαια, συμφωνώ και με την ε, πρόσφατη παρατήρηση, χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση ακριβώς γιατί είναι άκρος απαραίτητη και ουσιώδης και όχι μόνο για τη διαμόρφωση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης. Θα ήθελα όμως εδώ να υπενθυμίσω και να υπογραμμίσω κάποιες ε, πτυχές που κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητες. Στο έγγραφο επικοινωνίας της Κομισιόν προς τους ε, υπόλοιπους φορείς, την, Ευρω... την ε, Επιτροπή των Περιφερειών, την και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου στις 7 Ιουνίου, όπως θα έχουμε δει, στο κεφάλαιο 2 περιγράφεται η αξιολόγηση και οι συστάσεις της και γίνεται λόγος για τις επιπρόσθετες προσπάθειες που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι στα θέματα της απασχόλησης, της έρευνας και της ανάπτυξης, της ενεργειακής αποδοτικότητας, της τριτοβάθμιας παιδείας, εκπαίδευσης και της φτώχειας. Επιπλέον, ως επόμενα βήματα, στο ίδιο έγγραφο επικοινωνίας, γίνεται λόγος, και πρέπει αυτό να το υπογραμμίσουμε, πως τα κράτη-μέλη χρειάζεται να βρουν τρόπους για να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές επιπτώσεις των αλλαγών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και στο δελτίο τύπου της ίδιας μέρας της Κομισιόν για τις αναχώρα προτάσεις της πάνω στην ανάπτυξη και την απασχόληση γίνεται αναφορά ανάμεσα στα άλλα στην αγορά εργασίας και στην ανάγκη για την αύξηση της απασχόλησης. Ακόμη την καταπολέμηση της δομικής ανεργίας και τη μείωση της ανεργίας των νέων. Είναι θέματα που ξεκίνησε η Κομισιόν με την ετήσια έρευνα ανάπτυξης τον περασμένο Ιανουάριο και είναι φυσικό λόγω των εξελίξεων αυτή η έρευνα να διαφοροποιείται. Για τα θέματα αυτά θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ο Λάμπερτ Βαν Νίστερροϊ θέλει να μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ. Μερικές παρατηρήσεις για αυτή τη γνωμοδότηση. Ε, σε ψήφισμα του Κοινοβουλίου είπαμε ναι αρχικά για αυτή την στατική 2020, μετά για τη διακυβέρνηση και τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Και συμφωνώ απολύτως με αυτή τη σκέψη να το προωθήσουμε με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, για παράδειγμα στην Επιτροπή των Περιφερειών. Πρέπει να υπάρξει μια επίβλεψη αυτή τη πλατφόρμα 2020. Αρχικά υπάρχει η λήψη της απόφασης, μετά συγκεκριμένες ε, εμβληματικές πρωτοβουλίες και πολιτικές. Ε, αυτή είναι η δεύτερη φάση. Όμως εδώ βλέπω μια δήλωση της Επιτροπής των Περιφυρών, μια ανακοίνωση. Την πρώτη φορά αυτή η αξιολόγηση έγινε, αλλά ακροθυγός μάλλον. μετά για το... Λένε ότι δεν υπάρχει μια θετική ισορροπία, ένα θετικό ενεργητικό αν θέλετε, στον τρόπο με τον οποίο το χειρίστηκαν τα κάτι μελη Ουσιαστικά λέμε δηλαδή ότι αυτά που έκανε η Επιτροπή δεν ε, έφτασαν στο ύψος των προσδοκιών μας. Είναι κάτω από τις, ε, από τους, ε, τους στόχους μας. Αυτό που να πούμε λοιπόν. Αν θέλουμε να αλλάξουμε λοιπόν, πρέπει να πούμε από τώρα ότι θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Και μετά μπορεί η Επιτροπή Οικονομικών και Δημοσιονομικών Ζητημάτων να το εξετάσει εκ νέου. Πρέπει να πούμε δηλαδή ότι την επόμενη φορά πρέπει να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά να συμμετέσχει με πολύ πιο ενεργητικό ρόλο και ενεργό ρόλο και η Επιτροπή των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί προ το παρόν παίζουμε ένα πολύ περιφερειακό ρόλο και περιθωριακό ρόλο μάλιστα. Έχουμε θέσει στόχου στα τρία τέταρτα των δραστηριοτήτων να διεξάγονται σε τοπικό επιφερειακό επίπεδο. Προ το παρόν όμω αυτό δεν συμβαίνει και δεν είναι καθόλου ικανοποιητικά τα αποτελέσματα. Υπάρχουν περιφέρειες που δεν κάνουν ουσιαστικά τίποτα και μετά λαμβάνουν και φιλοφρονήσεις από την Επιτροπή ότι κάνετε το ένα, κάνετε το άλλο. Όμως ε, το θέμα είναι ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε μια πιο αυστηρή ε, στάση. Ο συνάδελφος έχει ήδη στοχεύσει σε αυτό, μόνος δεν χρειάζεται να υποβάλω τροπολογίες. Έτσι, Μιχαήλ. Προς αυτή την κατεύθυνση όμως κινούμε. Ευχαριστώ. Από ό,τι βλέπω δεν ζητά κάποιο άλλο το λόγο. Σπανίω λαμβάνω το λόγο. Ε, ο ρόλο μου είναι να διευκολύνω τη συζήτηση. Όμως θα ήθελα να πω δύο λόγια. Είναι μια καλή ευκαιρία, πιστεύω, να σημειώσουμε ένα γεγονός. Ένα στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να αποδεχόμαστε. Τα περισσότερα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά προγράμματα, ξεκινώντας με την ενιαία αγορά πριν μερικά χρόνια, τώρα για παράδειγμα με το εξάμεινο αυτό, ε, για την εισαγωγή μιας νέας προσέγγισης ε, στο συντονισμό των ε, πολιτικών συνοχής. Όλα αυτά τα προγράμματα δεν έχουν καμία... δεν εστιάζουν καθόλου, καθόλου στις περιφέρειες και στην διακυβέρνηση. Θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε περισσότερο στο τι προσφέρει αυτή η πολιτική ε, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη και στις αλλαγές. Αλλά και στο συντονισμό σε ό,τι αφορά την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση για την διαδικασία λήψη αποφάσεων. Θα πρέπει να το αναφέρουμε και για το θετικό στοιχείο και για το αρνητικό, δηλαδή και για τη συνεισφορά αλλά υπάρχουν και παράδειγμα και τα ζητήματα της ε, δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτή είναι η ερνητική πτυχή, που και αυτή μας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτές τις διαδικασίες. Βεβαίως, οι λύσεις ποικίλουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο περιθώριο ευελιξίας. Ωστόσο, θα πρέπει να αρχίσουμε να, συμμετέχουμε πιο ενεργά σε όλα τα μακροοικονομικά ζητήματα και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Γι' αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα που ανέλαβε αυτή την ε, πρόκληση ο συνάδελφος Μάικλ και έχουμε τώρα αυτή την ε, γνωμοδότηση. Αυτό όμως θα πρέπει να συνεχιστεί. Σήμερα λοιπόν το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποφασίσουμε την προθεσμή για την υποβολή τροπολογιών στις 22 λοιπόν αύριο μέχρι τις 6 το απόγευμα έχετε το περιθώριο. Α, Μίκαλ, βεβαίως και ήθελα να σου δώσω το λόγο. Αλλά ξέχασα, Μίκαλ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις συζητητές για τα σχόλιά τους. Είμαι εντελώ ανοιχτό. Αν θέλετε να ενισχύσουμε κάποιε θέσει και αν έχετε συγκεκριμένο κείμενο να προτείνετε, εγώ είμαι ανοιχτό και προσβλέπω σε κάτι τέτοιο. Ανέφερα την ολοκλήρωση την πολυεπιπεδική και θα ήθελα να υπάρχει και συμμετοχή, να ενταχθεί και συμμετοχή στο τοπικό επίπεδο στη διαδικασία. Ίσως όλοι μαζί να βρούμε καλύτερη διατύπωση. Ε, να είναι ισχυρότερη. Ας συνεργαστούμε λοιπόν. Και θα έχουμε καλύτερη δυνατότητα να ενισχύσουμε και την ε, περιφερειακή ανάπτυξη και την συνοχή. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Αν δεν υπάρχει τίποτα στα διάφορα στο 13, η επόμενη συνεδρίαση λαμβάνει η χώρα στις 11 και 12 Ιουλίου και θα είναι τελευταία συνεδρίαση πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Οπότε Λίγη συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ όσους μείνανε μέχρι τώρα μαζί μας. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας νύχτα.